Good afternoon, dear colleagues. Καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Καλώς ήρθατε στην παρουσίαση που θα μας κάνει ο πρόεδρος Εκτο ο κύριος Ντράγκη. Καλώς ορίστε και τον κύριο Ντράγκη μάλλον. Υιοθετούμε την ημερήσια διάταξη. Να σας ενημερώσω σχετικά με τις οργανικές ε, διαπραγματεύσεις. Αυτές αφορούν τον τριμερή διάλογο, το πεζικό πακέτο, το BRDS, REM, τον κανονισμό, δεύτερος τριμερής διάλογος, ε, διεξήχθη την 11η Σεπτεμβρίου. Συζητήσαμε το μορατόριο και διάφορα άλλα θέματα που μας απασχολούν. Ε, γιατί το Αμαρέλ και πώς τα ελέγχεται. Βάσει ενός εγγράφου ε, εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμφώνησαν οι υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μας δώσουν ένα έγγραφο με επιλογές προς συζήτηση στο μέλλον και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προβληματιστούν επί ενδεχομένων λύσεων για το άρθρο 32α προτείνει και το Κοινοβούλιο και τεχνικό έργο που έχει γίνει μέχρι τώρα ανεκρίθη και παρετάθη εντολή για να εξεταστούν και άλλες τάξεις το CR2, CR5 για τον διάλογο. Στι 12 Σεπτεμβρίου έγινε άλλο τριμερή διάλογο στο Στρασβούργο. Συζητήσαμε ε, μόχλευση, τα θέματα των κεφαλογικών μέσων, πυλώνα 2, μικροπροληπτικό πλαίσιο, ε, προσωρινή κάποια συμφωνία ίσως σε κάποια σημεία να επιτευχθεί, όμως οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν στον επόμενο τριμερή διάλογο που έχει προγραμματιστεί για τις 27 Σεπτεμβρίου του 2018. Και τώρα να καλωσορίσω εκ νέου τον κύριο Μάριο Ντράγκη για τον τρίτο διάλογο επινομισματικών ε, για το έτος 2018. Όπως γνωρίζετε, αυτός ο νομισματικός διάλογος λαμβάνει χώρα μετά από την τελευταία συναντήση του Διοικητικού Συμβουλίου που επιβεβαίωσε τη θέση του Ιουνίου της ΕΚΤ για τους προσανατολισμούς, για τα επιτόκια, για τη στεδιακή εξάλληψη των προγραμμάτων εξαγοράς ε, στοιχείων ενεργητικού και επενδυτική πολιτική ε, με κάποιες ρυθμίσεις νομισματικού χαρακτήρα, ευπρόσδεκτες οι αποφάσεις και θα συνεχίσουμε συζητώντας και την ανακοίνωση της ΕΚΤ τώρα που η νομισματική πολιτική δεν είναι και η πιο συνηθισμένη η ανακοίνωση της ΕΚΤ λοιπόν έγινε πολύ θετικά δεκτή από τις αγορές θα συζητήσουμε το θέμα δραστηριοτήτων των δανειοδοτικών των τραπεζών, τα θέματα ρευστότητας και άλλα ζητήματα, ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που πρέπει να παρακολουθούνται, κυρίως για τους κινδύνους και δεν βλέπουμε να υπάρχουν αρνητικές εξελίξεις μέχρι τώρα και αυτό ενισχύει τη θετική αξιολόγηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ντράγκη. Όλοι προσβλέπουμε στην επόμενη απόφαση. Οπότε θα ακούσουμε τι έχετε να μας πείτε και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής, κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι που είμαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μιλάω στην Επιτροπή σας. Πριν από 10 χρόνια η Ευρωζώνη μπήκε σε μια πολύ σοβαρή ύφεση και αυτή η κρίση εξέθεσε διαφορετικές αδυναμίες και υποχρεωθήκαμε να τις καλύψουμε. Δεν έχει ολοκληρωθεί η προσπάθεια ακόμα αλλά εμείς βλέπουμε τους καρπούς των προσπαθειών μας. Η ανάπτυξη υπήρχε θετική για περισσότερο από μια πενταετία και τα επίπεδα της ανεργίας είναι στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2008, συγκρίση με τον Νοέμβριο του 2008. Στα σχόλιά μου σήμερα θα συζητήσω την, το τρέχον περιβάλλον το οικονομικό και το ρόλο της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ σχετικά με τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος. Κατόπιν αιτήματος Επιτροπής σα. θα συζητήσω και την ανακοίνωση της ΕΚΤ που είναι αναπόσπαστο τμήμα τώρα πια της νομισματικής ε, πολιτικής. Λοιπόν, οι πληροφορίες διετέθησαν μετά την τελευταία μου επίσκεψη που έλαβε χώρα τον Ιούλιο και επιβεβαιώνει εν γέννη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της οικονομίας της Ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 0,4% στο δεύτερο τρίμηνο του 2018. Παρά κάποιες μειώσεις λόγω ε, των επιδόσεων του 2017 η οικονομία συνέχισε να παρουσιάζει ψηλά επίπεδα δυνατότητας χρήσεως των δυνατοτήτων. Ε, έχουμε τελικά προβλήματα ελλείψεως εργατικών χεριών σε κάποιους ε, τομείς ε, στην αγορά εργασίας και αυτό αντικατοπτρίζεται στα επίπεδα της ανεργίας στην Ευρωζώνη που ήταν στο 8,2% τον μήνα Ιούλιο έφτασε μια, το χαμηλότερο επίπεδο και πέντε χρόνια. Η απασχόληση όμως στην Ευρωζώνη τώρα έχει αυξηθεί κατά περίπου 9,2 εκατομμύρια λόγω της βελτίωσης κατά στην αγορά εργασίας και των γενικότερων συνθήκων. Τα νοικοκυριά έχουν διαθέσιμο εισόδημα που αυξάνεται με τις υψηλότερους ρυθμούς που είδαμε τελευταία δεκαετία μεγαλύτερο εισόδημα προωθεί την κατανάλωση που αναμένεται να πτυχθεί κατά 1,5% το έτος 2018. Αυτοί οι παράγοντες μαζί με τις επιχειρηματικές επενδύσεις που τονώζονται από το ευνο, ευνοϊκές συνθήκες και τα κέρδη των επιχειρήσεων και τη ζήτηση, όλα αυτά υποστηρίζουν την ανάπτυξη. Τώρα βλέποντας τι θα γίνει στο μέλλον, οι, οι μακροοικονομικές προβολές του προσωπικού μας δείχνουν ότι θα έχουμε συνεχιζόμενη ευρή ανάπτυξη της οικονομίας Ευρωζώνης. Μέσα ετήσια ανάπτυξη προβλέπεται να είναι 2% το 2018, 1,8% το 2019 και 1,7% το 2020 με μια μείωση πολύ μικρή ε, το 2018 και 2019 που αυτό θα την κατοπτρίζει μεγαλύτερο, πιο αδύναμο παγκόσμιο εμπόριο οι κίνδυνοι που περιβάλλουν την Ευρωζώνη μπορεί να θεωρηθούν ότι τελικά είναι εξισορροπημένοι παρόλο που η απειλή του προστατευτισμού, ε, οι ευάλωτες αναδυόμενες αγορές και οι μεταβλητός χαρακτήρας χρηματοστατικών αγορών δημιουργούν κάποια προβλήματα. Οι φορολογικές πολιτικές σε κάποιες χώρες της Ευρωζώνης ίσως να είναι λιγότερο ουδέτερες από ό,τι περιμέναμε πριν από λίγο. Όσον αφορά τον πληθωρισμό, ο πληθωρισμό HICP ήταν 2% τον Αύγουστο, μειώθηκε το 2,1% τον Ιούλιο. Ε, τελικά ο μέσος όρος του πληθωρισμού είναι ψηλότερο από το πρώτο μήνες του έτους και αντικατοπτρίζει τη μεγάλη αύξηση της τιμής του πετρελαίου. Αν δούμε τώρα τι γίνεται με τον υποβόσκοντα πληθωρισμό, βλέπουμε ότι είναι χαμηλός, αλλά έχει αυξηθεί σχετικά με το παρελθόν, διότι υπάρχουν μεγαλύτερε πιέσει όσον αφορά τις εσωτερικές ε, τιμές. Ε, ο υποβασκο πληθωρισμός θα αυξηθεί περαιτέρω του επόμενου μήνε διότι τελικά η έλλειψη εργατικών ε, χεριών στην αγορά εργασία οδηγεί σε αύξηση των αμοιβών. Παραδείγματο χάρη, η ετήσια ανάπτυξη όσον αφορά τα ημερομίστια στο, στην Ευρωζώνη αυξήθηκε από ένα 5% το 2017 σε 1,7% ε, το πρώτο τρίμηνο του 2018 και 2,2% το δεύτερο τρίμηνο. Αυτό στηρίζει την πεποίθησή μας ότι η αύξηση των αμοιβών θα συνεχιστεί, όπως οι συμφωνίες περιμεριστίων πολύ συχνά έχουν διάρκεια δύο έτη περισσότερα. Βλέποντα τι θα γίνει τόσο στο μέλλον, τα ετήσια επίπεδα του πληθωρισμού θα είναι περίπου στα παρόντα επίπεδα του επόμενου μήνε και προβλέπεται ότι θα φτάσουν 1,7% κάθε έτος από την, περίοδο από τώρα μέχρι το 2020. Αυτός ο σταθερός ρυθμός δείχνει μια μειούμενη συνεισφορά από τους μου βασικούς συντελεστές του γενικού δίκτου και σχετική αύξηση του υποβόσκοντα πληθωρισμού. Ε, αυτή τη δυναμική, οι προβλέψεις της ΕΚΤ προβλέπουν ε, ότι ο πληθωρισμός εκτός από τρόφιμα και ενέργεια θα φτάσει το 1,8% το 2020. Τώρα, εν γέννη, οι πρόσφατες εξελίξεις δικαιώνουν τι πρώτερε αξιολογήσει του Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά το μεσοπρόθεσμο πληθωρισμό, τι προβλέψει περί αυτού. Και στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικό Συμβουλίου αποφάσισε να διατηρήσει τη σημαντική εθνομισματική πολιτική, την τόνωση μέσω νομισματικής πολιτική στην παρούσα μορφή, σύμφωνα με το προσωρινό σχέδιο που ανακοινώθηκε στην συνέντευξη τύπου τον Ιούνιο στη Ρήγα να μειωθεί ο μηνιαίο αριθμός της αγοράς στοιχείων ενεργητικού σε 15 εκατομμύρια δισεκατομμύρια τον Οκτώβριο μέχρι το τέλος του έτους. Και προβλέπουμε ότι με επιφύλαξη των στοιχείων που επιβεβαιώσουν την πρόβλεψή μας θα σταματήσουμε αυτές τις αγορές. Αυτό δεν σημαίνει ότι η νομισματική πολιτική μας δεν θα είναι ευέλικτη για τις βασικές μας προσδοκίες για την αύξηση του πληθωρισμού. Για να αυξηθεί ο πληθωρισμός πραγματικά πρέπει να παραμείνουμε υπομονετικοί, συνετοί και ε, ε, επίμονοι σταθμίζοντας ε, την νομισματική μας πολιτική. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση θα συνεχίσουμε να παρέχουμε σημαντική νομισματική τόνωση συνδυάζοντα τρία μέτρα πολιτικής. Πρώτα απ' όλα θα δίνουμε αυξημένους προσανατολισμούς όσον αφορά τα επιτόκια τα βασικά της ΕΚΤ που περιμένουν να παραμείνουν στα παρόντα επίπεδα τουλάχιστον κατά τη διάρκεια του θέρους του επόμενου έτους και εν πάση περιπτώσει στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να εξασφαλίζεται η συνεχή σύγκληση του πληθωρισμού προς το στόχο μας. Δεύτερον, ε, λοιπόν, οι αγορές αξιογράφων στοιχείων εργητικού που θα κάνουμε μέχρι το τέλος του έτους θα συνεχιστούν και τρίτον, οι επανεπενδύσεις ε, του αποθέματος ε, των αποκτημένων ε, αξιογράφων. Η νομισματική μας πολιτική και τα μέτρα αυτής συνέβαλαν τα μάλα στη θετική οικονομική εξέλιξη στην Ευρωζώνη. Εάν θεωρήσουμε ότι όλα τα μέτρα της πολιτικής που ελήφθησαν από τα μέσα του 2014 οι εκτιμήσει του προσωπικού δείχνουν ότι γενικό αντίκτυπο στην Ευρωζώνη και στο ΑΕΠ, στην ανάπτυξη του ΑΕΠ και τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη και σε δύο περιπτώσεις είναι στο 1,9% σορευτικά στην περίοδο 2016 μέχρι 2020. Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της επικοινωνίας της ε, Κεντρικής Τράπεζας που προτείνατε για την σημερινή μας ε, συνεδρίαση για το θέμα αυτό. Πράγματι, οι κατευθύνσει για το μέλλον είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσο για όλε τι κεντρικέ τράπεζε, καθώ ε, τα συμβατικά μέσα πλέον έχουν φτάσει, τα συμβατικά νομισματικά μέσα έχουν φτάσει στο κατώτατο όριο και η ΕΚΤ δεν αποτελεί εξαίρεση. Οπότε, οι κατευθύνσει ε, που δίνουμε για το μέλλον έχουν εξελιχθεί από όταν ξεκινήσαμε τον Ιούλιο του 2013. Χοντρικά μιλώντας, έχουν περάσει από τρεις όταν ε, ξεκινήσαμε το 2013, στόχος μας ήταν ε, να προσπαθήσουμε να σταθεροποιήσουμε τις νομισματικές ε, συνθήκες της Ευρωζώνης και ειδικά το θέμα των επιτοκίων στις χρηματαγορές από την υψηλή κινητικότητα που προέκυψε από τις αμερικάνικες αγορές ως αποτέλεσμα του επεισοδίου τον Μάιο-Ιούνιο 2013 κατά την διάρκεια της ε, δεύτερης ε, φάσης. Η κατεύθυνση που δώσαμε στόχο είχε ακριβώς να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των ε, αγορών στοιχείων ενεργητικού, τις οποίες κάναμε. Εκφράζοντας τις προσδοκίες του Διοικητικού Συμβουλίου για την μελλοντική πιθανή πορεία των επιτοκίων, διασφαλίζαμε ότι ο αντίκτυπος των αγορών στις μακροχρόνιες αποδόσεις δεν θα εξουδετερώνονταν από τις προσδοκίε των αγορών για βραχυπρόθεσμη αύξηση των επιτοκίων. Από τον Ιούνιο του 2018 έχουμε εκφράσει την προσδοκία μας ότι υπό την αίρεση των δεδομένων που θα επιβεβαιώνουν την πρόβλεψή μας για τον μεσοπρόθεσμο πληθωρισμό, οι αγορές αυτές θα σταματήσουν μετά τον Δεκέμβριο του 2018. Καθώς ε, είχαμε εδώ και καιρό συνδέσει τον ορίζοντα για τα επιτόκια με το τέλος των αγορών ε, αυτών και είχαμε δώσει τις ανάλογες ενδείξεις, η ανακοίνωση ενός ε, σχεδίου υπό όρους ε, σημαίνει ότι θα πρέπει να ξαναρχίσουμε να δίνουμε μια κατεύθυνση για το πώς θα κινηθούν τα επιτόκια. Το να κατευθύνουμε δηλαδή τις προσδοκίες αυτές είχε μεγάλη σημασία γιατί η πορεία του πληθωρισμού θεωρούσαμε ότι πήγαινε και εξακολουθεί να είναι υπό την αίρεση μιας δομής επιτοκίων που θα αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες των συνεχών αλλαγών επιτοκίων για μια εκτεταμένη περίοδο μετά το Δεκέμβριο του 2018. Ήταν σημαντικό λοιπόν για εμάς να διατηρήσουμε έλεγχο επί των μήνυμάτων που εξυπονοούνται στις ανακοινώσεις μας για την νομισματική πολιτική. Σε αυτή την κρίσιμη καμπή έπρεπε να διαβεβαιώσουμε τους επενδυτές ε, και το κοινό ότι η αλλαγή αυτή στις αγορές οποίες έκανε η τράπεζα δεν θα εμπόδιζε την ανάπτυξη και την ομαλοποίηση του πληθωρισμού έχοντας αυτά κατά νου. Τον Ιούνιο του 2018 είπαμε ότι αναμέναμε τα επιτόκια να παραμείνουν στο τωρινό επίπεδο τουλάχιστον για ολόκληρο το καλοκαίρι του 2019 και σε κάθε περίπτωση για όσο απαιτείται έτσι ώστε ο πληθωρισμός να ευθυγραμμίζεται με τις προσδοκίες μας για μία βιώσιμη πορεία προσαρμογής. Οι κατευθύνσεις αυτές, τις οποίες επαναλάβουμε και τον Ιούλιο φέτος και αυτόν τον μήνα, περιέχει δύο μέρη. Το πρώτο είναι μέχρι και το καλοκαίρι του 2019 μία διατύπωση η οποία μας λέει πότε αναμένουμε κάποιες συνθήκες οι οποίες θα μας οδηγούσαν σε μία πρώτη αύξηση των επιτοκίων και δεύτερον ένα στοιχείο που εξαρτάται από τα κράτη και δείχνει ότι θεωρούμε ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν σταθερά για όσο απαιτείται για να συνεχιστεί η απαραίτητη σύγκληση του πληθωρισμού σε επίπεδα που είναι κάτω αλλά κοντά στο 2% μεσοπρόθεσμα. Όπως αποδείχτηκε η ευθυγράμμιση των προσδοκιών της αγοράς με αυτόν του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν άμεση και ήπια. Η νέα διατύπωση βοήθησε τους συμμετέχοντες στις αγορές να αντιληφθούν καλύτερα την αντίδρασή μας και να προσαρμόσουν τις προσδοκίες τους ανάλογα. Βεβαίως, η κατεύθυνση των ε, συνθήκων αυτών μέσω των ενδείξεων που δίνουμε στους επαγγελματίες ε, των αγορών είναι μόνο μέρος των ε, καθηκόντων μας. Είμαστε υπεύθυνοι για τη σταθερότητα τιμών για τα 340 εκατομμύρια ανθρώπους της Ευρωζώνης και βεβαίως έχει μεγάλη σημασία να έχουμε και την εμπιστοσύνη των πολιτών ως κεντρική τράπεζα και για την καταλληλότητα των πολιτικών μας και για τον σκοπό αυτό έχουν κέρια σημασία οι ακροάσεις ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί έτσι μπορούμε να εξηγούμε τους λόγους για τις αποφάσεις μας και πώς επηρεάζουν τις ζωές των ανθρώπων. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με βάση το πλαίσιο που έχει διαμορφώσει το πρωτογενές δίκαιο έχουν ανταποκριθεί στην ανάγκη για σοβαρότερη και ισχυρότερη διαφάνεια και ένα μεγαλύτερο βαθμό λογοδοσίας που προέκυψε κατά τη διάρκεια της κρίσης. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να επαναπαυθούμε. Γνωρίζουμε ότι η διατήρηση της εμπιστοσύνης προς την ΕΚΤ σημαίνει ότι πρέπει να επαγρυπνούμε. Και βεβαίω αντιμετωπίζουμε σοβαρέ προκλήσει. Παραδείγματο χάρη από τον Ιανουάριο του 2015, η ΕΚΤ δημοσιεύει τακτικά τις αποφάσεις ε, του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν την νομισματική πολιτική. Και όπως ε, αποδεικνύουν και οι συζητήσεις που έχουμε κάνει εντός αυτής της ε, αιθούσης, αυτές οι πληροφορίες σας δίνουν την δυνατότητα σε εσά και σε όποιον άλλο ενδιαφέρεται να εξετάσει σε μεγαλύτερο βάθος την πολιτική της ΕΚΤ. Ταυτόχρονα Βεβαίω ε, έχουμε έτσι την ευκαιρία και εμεί να εξηγήσουμε τι αποφάσει μα και να αποδείξουμε ότι δρούμε σύμφωνα με την δημοκρατική εντολή μα. Τα τελευταία χρόνια επίση έχουμε εντείνει τι προσπάθειέ μα ε, στον τομέα τη επικοινωνία. Έχουμε έρθει σε επαφή με πολίτε σε 19 χώρε που βεβαίως έχουν διαφορετικές προσδοκίες από την ΕΚΤ. Έτσι έχουμε ενισχύσει την πολιτική επικοινωνία και απευθυνόμαστε απευθείας σε ένα ευρύτερο ακροατήριο. Πέρα από τις θεσμικές μας δραστηριότητες, οι συνάδελφοί μου στο Εκτελεστικό Συμβούλιο έχουμε λάβει μέρος σε 180 εκδηλώσεις τα τελευταία δύο χρόνια, το 1 τέταρτο από αυτές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αν περιλάβω δε και τα think tank ιδρύματα μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ε, και κρατικούς ε, φορείς. Έχουμε βγάλει περισσότερες λόγους σε αυτά τα φόρα παρά στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες. Τα μέλη της ε, τράπεζας έχουν συμπληρώσει αυτή την προσπάθεια με ένα πρόγραμμα επαφών που στόχο έχει ακριβώς τα τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα πανεπιστήμια και εξηγεί τον ρόλο της ε, Κεντρικής Τράπεζας και το πώς προσπαθεί να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση. Το ίδιο κάνουμε και στην ιστοσελίδα μας που τώρα έχει βίντεο επεξηγηματικά και πίνακες που περιγράφουν περίπλοκα ζητήματα με έναν τρόπο πιο απλό. Έχουμε αρχίσει να χρησιμοποιούμε νέα μέσα όπως το YouTube, το LinkedIn και το Twitter όπου έχουμε σχεδόν 400.000 ακολούθους. Να καταλήξω λοιπόν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο εκπροσωπεί του πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, είναι ακριβώ αυτό το οποίο θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και κατανόηση των αποφάσεων τη ΕΚΤ. Και υπ' αυτήν την έννοια συνεισφέρει στην αποτελεσματικότητα τη νομισματική πολιτική όμω η συνεισφορά σα δεν τελειώνει εδώ. Ω συνομοθέτες έχετε έναν ρόλο να παίξετε έτσι ώστε η Ευρώπη να είναι προετοιμασμένη για του κινδύνου που ανέφερα στην εισαγωγή μου εάν αυτοί υλοποιηθούν έχουμε δει ότι πέρα αντί να βλάπτει την ε, ανάπτυξη, ένα ισχυρό ρυθμιστικό πλαίσιο έχει μεγάλη σημασία για να διασφαλίσουμε μια ισχυρή μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Σήμερα, 10 χρόνια μετά την αρχή της οικονομικής κρίσης, υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει όσον αφορά το νομοθετικό πλαίσιο. Και καθώς πλησιάζουμε στο τέλος αυτής της ε, νομοθετικής θητείας, πρέπει ακριβώς να ατράξουμε αυτή την ευκαιρία. Γι' αυτό αναμένω την στήριξή σας για να διαμορφώσουμε το πλαίσιο το οποίο θα παρέχει την απαραίτητη σταθερότητα στις αγορές, προστατεύοντας έτσι τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εργαζόμενους και φορολογούμενους. Σας ευχαριστώ. Είμαι στην διάθεσή σας για ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ντράγκη για τις παρατηρήσεις που κάνατε και κυρίω για τα όσα είπατε για τη σημασία του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μια και είμαστε ένα βήμα που προκρίνει την διαφάνεια σε σχέση με θέματα πολιτικής της ΕΚΤ. Και βέβαια είμαστε και ο συνομοθέτης και μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως εμείς θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε έτσι ώστε να κλείσουμε όσο το δυνατόν πιο πολλά από τα από τις νομοθετικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στα πλαίσια της τρέχουσας θητείας ή έτσι ώστε να βελτιωθεί το νομοθετικό πλαίσιο υπέρ της οικονομικής σταθερότητας και με στόχο να συμπληρώσουμε και την Τραπεζική Ένωση στα πλαίσια της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Ο Μάρκους Φέρμπερ από το ΕΛΚ είναι ο πρώτος ομιλητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Διοικητά. Και από μένα σας ε, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις δηλώσεις σας. Αναπτύξατε ένα θετικό σενάριο για τις οικονομικές εξελίξεις, όμως από ό,τι φαίνεται έχουμε τα πρώτα νέα σύννεφα που μαζεύονται, κάποια από αυτά τα σύννεφα τα έχουμε και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, το τελευταίο Σαββατοκύριακο στην Σύνοδο Κορυφής είχαμε το θέμα του εάν τελικά θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο ή όχι. Βεβαίως αυτό επηρεάζει και την ε, δική σας ε, την δουλειά. Αν και το Ηνωμένο Βασίλειο βεβαίως ε, δεν υιοθέτησε ούτε είχε ποτέ την πρόθεση να υιοθετήσει το ευρώ όμως το ερώτημά μου είναι το εξής. Πώς προετοιμάζεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την περίπτωση ενός σκληρού Brexit για τις ε, πιθανές αναταράξεις των αγορών. Υπάρχει κάτι, υπάρχουν κάποιες συνεννοήσεις με την Τράπεζα της Αγγλίας. Πώς βλέπετε την μελλοντική συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο στον νομισματικό τομέα και στην περίπτωση και ενός έφτακτου Brexit τίθεται το ερώτημα επίσης της μελλοντική συνεργασίας με την Τράπεζα της Αγγλίας, ειδικά όσον αφορά την επιτήρηση του Euroclearing και την ε, παροχή ρευστότητα σε περιπτώσεις ανάγκης. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μας κάνετε μια παρουσίαση αυτών των ρυθμίσεων. Uh, thank you. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να μιλήσω για τις απραγματεύσεις που τρέχουν, αλλά να σας υπενθυμίσω πως η ΕΚΤ δεν αποτελεί τμήμα των διαπραγματευτών. Οπότε εμείς αναμένουμε τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης πριν αποφασίσουμε ποια θα είναι η επόμενη πορεία που θα ακολουθήσουμε. Προφανέστατα θα θέλαμε οποιαδήποτε λύση να μην υποσκάψει την συνοχή της ενιαίας αγοράς. Όμως Ξέρετε κι εσείς πως έχουμε συστήσει μια ομάδα εργασία με την Τράπεζα της Αγγλίας και αυτή τη στιγμή εξετάζουμε διάφορα σενάρια ε, που θα μπορούσε ε, ενδεχομένως να, στα οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να καταλήξει η διαπραγμάτευση, αλλά δεν γνωρίζουμε ποιο θα είναι τελικά αυτό το οποίο θα επιλέξουμε. Εμείς έχουμε κάνει κάποιους υπολογισμούς και βλέπουμε πως ε, ε, οι επιπτώσεις αθρηστικά θα είναι αρκετά μετρημένες ε, και σε χρηματοπιστωτικό επίπεδο νομίζουμε ότι η μοναδική εξαίρεση που θα είναι σημαντική ε, για το clearance είναι η περίπτωση που θα έχουμε ένα σκληρό Brexit ε, της ε, χειρότερης ε, πιθανών έκβασης και εκεί σε κάποιο επίπεδο το clearing ε, το οποίο αυτή τη στιγμή αποτελείται από πολυεπίπεδες συμβάσεις θα επηρεαστεί. Αυτό είναι άγνωστο. Αλλά σε γενικές γραμμές η συνεργασία με την Τράπεζα της Αγγλίας είναι καλή. Αλλά επαναλαμβάνω, όλα αυτά θα εξαρτηθούν από το τελικό αποτέλεσμα των διαπραγματευσεων Φόλο Follow-up ερώτηση παρακαλώ. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή συνίσταται σε επιχειρήσεις να προετοιμαστούν για την χειρότερη περίπτωση, γιατί το περιθώριο είναι πάρα πολύ σύντομο, εάν ε, υπάρξει τελικά μια συμφωνία έχετε και καταρτήσει κι εσείς ένα σενάριο για την χειρότερη των περιπτώσεων εντός της ΕΚΤ. Εκτός μικροφώνου. Final Σας είπα, εμείς θα περιμένουμε να δούμε ποιο είναι το, τελευταίο, το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό που έχουμε ζητήσει από όλους τους εμπλεκόμενους να κάνουν όλες τις προετοιμασίες, αλλά δεν έχουμε λάβει καμία απόφαση και δεν έχουμε καμία δέσμευση για να γνωρίζουμε τι θα κάνουν οι δημόσιες αρχές. Γιατί αυτό αποτελεί κομμάτι κομβικό της τελικής διαπραγμάτευσης και σας επαναλαμβάνω, εμείς στις διαπραγματεύσεις δεν συμμετέχουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και βεβαίως παροτρύνουμε όλους να έχουν κάποιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης, παρόλο που εμείς θέλουμε να περάσει το σενάριο το βασικό, που είναι μια θετική και λογική συμφωνία, κάτι το οποίο θεωρούμε πως ακόμα γίνεται. Υπερβάος Περές, ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ που απαντήσατε σε ερωτήσεις ε, που σας έχουμε κάνει, αλλά είναι δύο σημεία στα οποία θα ήθελα να σταθώ. Καταρχήν, μετά την πρώτη ανταλλαγή απόψεων που κάναμε όταν είχατε έρθει την προηγούμενη φορά στην Επιτροπή μας, είχαμε δει για την Τράπεζα της Λετωνίας πως ενδεχομένως θα υπάρξει μια δυσκολία ε, λόγω της ε, νομιμότητας του ε, Προέδρου της Κεντρικής, ε, του, της Κεντρικής Τράπεζας γιατί η κυβέρνηση είχε ζητήσει να πάυσει από τα καθήκοντά του. Και αυτό βέβαια επηρεάζει και το ολόκληρο περιβάλλον και τη διακυβέρνηση του ευρωπαϊκού ε, συστήματος και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα ήθελα να μου πείτε λοιπόν υπάρχει κάποιο νομικό κενό το οποίο θα πρέπει να καλύψουμε και θα μπορούσε η ΕΚΤ να γνωρίζει όταν υπάρχουν ε, ε, δυσκολίες για παράδειγμα με μία εθνική κεντρική τράπεζα. Και επίσης την περασμένη εβδομάδα στο Βερολίνο ε, βγάλατε ένα λόγο και μιλήσατε για την ανάγκη σταθεροποίησης στις οικονομίες της Ευρωζώνης. Πιστεύετε λοιπόν πως οι προτάσεις που είναι υπό διαπραγμάτευση μετά από πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι χρήσιμες, ακολουθούν τη σωστή κατεύθυνση. Πιστεύετε πως είναι θέμα ε, του Συμβουλίου να κάνει μια προσπάθεια ακόμα έτσι τουλάχιστον μέχρι τη θητεία μας αυτές οι προτάσεις να έχουν ε, προχωρήσει για να δούμε αν μπορούμε και εμείς τις προτάσεις αυτές να προσθέσουμε κάτι. Για το πρώτο, για το πρώτο θέμα, για το τι θα γίνει με τα θέματα ε, με την νομοθεσία για, για το ξέπλυμα χρήματος, εντάξει. Είναι δεδομένο ότι η κατάσταση σήμερα δεν είναι ικανοποιητική. Και αυτό που κάνει η ΕΚΤ σήμερα είναι να είναι σε μια ομάδα εργασίας που έστησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε πρώτα απ' όλα να έχουμε καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών κατά του ξεπλήματος και των εποπτικών αρχών στο θέμα αυτό, και να σας πω ότι βέβαια δεν κλείνει εκεί το θέμα. Δηλαδή κάποιες πληροφορίες θα πρέπει να τις μαθαίνουν όλοι οι απόπτες και να κυκλοφορούν και σε όλες τις σχετικές αρχές. Η θέση της ΕΚΤ είναι πως θα έπρεπε, και νομίζω το ίδιο ακούσατε ε, γιατί το είπε και η Ντανιέλ Νουή, ότι χρειάζεται μία αρχή κατά της νομιμοποίησης του παράμονου χρήματος που θα είναι πανευρωπαϊκή. Δηλαδή, όχι μόνο εθνικά, όχι μόνο στη ζώνη ευρώ, αλλά και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν τω μεταξύ, εμεί έχουμε δημιουργήσει και αυτή τη στιγμή ενισχύουμε ε, μία πύλη, πύλη εισόδου, έτσι ώστε τα θέματα ε, ξεπλήματος να τα βλέπουν οι εποπτικές αρχές μαζί με το τμήμα ε, το δικαστικό της, της ΕΚΤ. Θυμηθείτε όμως πως η ΕΚΤ δεν είναι αρμόδια για την ε, πρόληψη και για την επιβολή της νομοθεσίας για την ε, νομιμοποίηση παράνομου χρήματος. Και δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε και πάρα πολλά για να αλλάξουμε την κατάσταση. Εδώ πρέπει να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν για να γίνει κάτι. Και για τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με τη σταθεροποίηση και σχετικά καθήκοντα. Ήσασταν πολύ ευγενικοί που μιλήσατε για τη δήλωση που έκανα στο Βερολίνο, αλλά εγώ δεν μπαίνω σε λεπτομέρειε των διαφόρων προτάσεων. Έχουμε αρκετέ προτάσει στο τραπέζι και κάθε μία σε κάποιο βαθμό έχει θετικά στοιχεία. Αλλά βέβαια έχει και σημεία περίπλοκα δυσκολίες. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολο ακόμα να επιλέξουμε μία από τις πολλές αυτές προτάσεις. Οποιαδήποτε πρόταση στο χώρο αυτό θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον δύο χαρακτηριστικά. Δηλαδή, επαρκής έτσι ώστε να επιτυγχάνει τη σταθεροποίηση. Και τι σημαίνει επαρκής. Και δεύτερον, η εμβέλεια. Σε αυτό θα προσθέσω ότι δεν θα πρέπει να στρεβλώνει και τα κίνητρα που έχουν τα κράτη-μέλη να αλαμβάνουν από, ε, αποφάσεις για την νομισματική τους πολιτική που δεν θα είναι επικίνδυνες. Δηλαδή να μην υπάρχει τόσο ηθικός κίνδυνος. Όταν λέμε λοιπόν επαρκής αν δείτε πώς αποδίδει στην νομισματική ένωση που είναι πιο προχωρημένη από τη δική μας η σταθεροποίηση, θα δείτε πως η κατανομή κινδύνου σε μεγάλο βαθμό, που είναι απαραίτητο για να αντιμετωπίσει τα διάφορα σοκ, αναλαμβάνεται από τον ιδιωτικό κλάδο. Και γιατί, γιατί αυτές οι νομισματικές ενώσεις έχουν πολύ ανεπτυγμένες και αγορές κεφαλαίων και τραπεζικές ενώσεις. Το δημόσιο κομμάτι λοιπόν είναι καλά πλαισιωμένο. Οπότε το πρώτο συμπέρασμα είναι πως το μέγεθος αυτής της δημοσιονομικής σταθεροποίησης και η σχετική αυτή λειτουργία ε, μειώνεται όσο μεγαλώνουν η Τραπεζική Ένωση και η Νομισματική Ένωση. Και το αντίστροφο. Αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να μην κάνουμε τίποτα. Ούτε για την αγορά κεφαλαίων, ούτε για την Τραπεζική Ένωση, ούτε για το κομμάτι της σταθεροποίησης. Αυτό το αποκλείουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μπέρτ Καλημέρα σας κύριε Ντράγκη, θα μιλήσω γερμανικά. Κύριε Ντράγκη, λάβατε μία επιστολή από τον Καλημέρα σας. Λάβατε μία επιστολή από τον ε, Ιταλό Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, ε, τον Σαβόνα, ο οποίος παρουσιάζει κάποιες ιδέες του για τον αναγκαίο μετασχηματισμό της Ευρωζώνης. Και βεβαίως αυτό συνδέεται και με την ε, δική μου την παρατήρηση ότι η Ευρωζώνη δεν αποτελεί μία ιδανική ζώνη νομίσματος. Ε, λοιπόν, και βεβαίως από τις ε, προθέσεις της ε, Ιταλικής κυβέρνησης αυξάνονται και οι ανησυχίες ε, αλλού στη Γερμανία το τι γίνεται με τις απαιτήσει target που είναι στο ύψος των χιλίων δισεκατομμυρίων ευρώ. Τι θα γίνει με αυτές στην περίπτωση στην οποία αποχωρήσει μονομερός μια χώρα η οποία έχει χρωστούμενα στον μηχανισμό target. Γνωρίζω ότι νομικός ε, δεν είναι δυνατόν, αλλά μπορεί να, γνωρί, να αγνοήσει τη νομική βάση η Ιταλία. Και υπάρχουν βεβαίως και δύο πρώην συναδελφοί μας εδώ πέρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που τώρα έχουν γίνει υπουργοί της κυβέρνησης ε, και είχαν πει ότι στην περίπτωση αυτή θα έπρεπε η Ιταλία να αποπληρώσει τα χρέη της. Αλλά αυτό, εξ όσων γνωρίζω, δεν έχει κάποια νομική βάση. Στην κατεύθυνση που δίνετε την μελλοντική θα ε, στείλετε και κάποιο μήνυμα για το τι θα γίνει με τις απαιτήσει ε, του μηχανισμού Target σε περίπτωση μονομερούς αποχώρησης μια χώρα από τον μηχανισμό και μια σχετική ερώτηση. Δεν θα ήταν δυνατόν το σύστημα αυτό να διαμορφωθεί έτσι ώστε οι υποχρεώσει στο μηχανισμό αυτό να γίνουν χρέο των κεντρικών τραπεζών έτσι ώστε να υπάρχει μία νομική βάση με κάποιο μεταβλητό επιτόκιο να μιμείτε τον τωρινό μηχανισμό αλλά με την σαφή πρόβλεψη ότι σε περίπτωση αποχώρησης ε, μιας χώρας από την Ευρωζώνη είναι και πληρωτέο αυτό το χρέος. my sense... Κοιτάξτε, τι πιστεύω. Καταρχάς το θέμα που θέσατε είναι τουλάχιστον περιπλοκότατο νομικό. Το λιγότερο μπορούμε να πούμε και δεν είναι στα χέρια τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να το διευθετήσει. Το δεύτερο τμήμα τη απαντήσεώ μου είναι το εξή. Οποιοδήποτε προσδιορισμό για τον στόχο 2, είτε ρητό είτε υπονοούμενο, θα καταστρέψει την νομισματική ένωση. Ο στόχο 2 είναι ένα σύστημα πληρωμών. Συνεπώ, αν αρχίσουμε να περιορίζουμε το ποσό των πληρωμών που μπορούν να πραγματοποιούν οι πολίτε, καταστρέφουμε την ένωση πρότεινα αυτό, λέει ο κύριος Λούκε. Sorry, Mr. You first... Και κύριε Λούκε, συγγνώμη, αφήστε τον να ολοκληρώσει και μετά, αν υπάρχει χρόνο, θα κάνετε για άλλη ερώτηση. I think I have... Κοιτάξτε, ολοκλήρωσε, λέει ο κύριος Ντράγκη. Νομίζω τελείωσα. I, I have not... Κοιτάξτε, δεν διατηνόμουν κάτι τέτοιο. Δεν είπα να περιοριστούν οι λειτουργίες του συστήματος του στόχου. Τι πρότεινα εγώ. Ότι οι θέσεις των στόχων ίσως να μετατραπούν σε μέσα χρεών να μετατραπούν σε μέσα χρεών, ούτως ώστε οι εθνικές κεντρικές τράπεζες, η Εθνική Κεντρική Τράπεζα που έχει αυτούς τους στόχους χρεών, να είναι νομικά υπεύθυνη για αποπληρωμή του χρέου σε περίπτωση εξόδου από το ευρωσύστημα. Δεν σχετίζεται καθόλου με τη λειτουργία του συστήματος στόχων όταν όλοι είναι εντός του συστήματος του ευρωπαϊκού. Σε περίπτωση εξόδου πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για την πιθανότητα μια κυβέρνηση να μην είναι πρόθυμη να εξυπηρετήσει τους στόχους ε, του συστήματος. Τις θέσεις στόχους. Απάντηση. Κατά κάποια έννοια έτσι έχουν τα πράγματα. Διότι η εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής είναι αποκεντρωμένη και υπάρχουν εγγυήσεις έναντι αυτών των θέσεων. Αυτή είναι η παρούσα κατάσταση το νομικό έδαφος, νομική βάση. Θεωρώ ότι είναι κάτι αδύνατο. Μιλάμε για μια αδύνατον να υπάρξει υπόθεση. Αδύνατον συμβεί. Αλλά η νομική θέση είναι αρκετά σαφή, Υπάρχει. Για να αλλάξουν τα πράγματα και να μετατροπούν αυτές οι ευθύνες, αυτές οι υποχρεώσεις ε, και να γίνουν κεντρικές ευθύνες της ΕΚΤ, δεν προβλέπονται από το παρόν πλαίσιο της νομισματικής πολιτικής το καταστατικό της ΕΚ δεν προβλέπει κάτι τέτοιο. Προβλέπουμε αποκεντρωμένη εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής. Ευχαριστώ. Thank you very much. Uh, Thank you, Ευχαριστώ, λέει κυρία Μπίρνη. Μετά την ομιλία για την κατάσταση στην Ένωση του κυρίου Γιούνκερ και η δυνατότητα το ευρώ να γίνει διεθνές αποθεματικό νόμισμα, ποιες είναι οι στρατηγικές τα στατηγικά ωφέλη, μειονεκτήματα να επιτευχθεί αυτό εν συγκρίση με την παρούσα κατάσταση. Ποια συγκεκριμένα βήματα απαιτείται να γίνουν για να το πετύχουμε αυτό και ποιο ρόλο μπορεί να παίξει η ΕΚΤ να αυξήσει τη θέση του ευρώ ε, στο παγκόσμιο προσκήνιο. Σας ευχαριστώ. Απάντηση. Κοιτάξτε. Ευχαριστώ. Να πω πρώτα απ' όλα ότι η πρόθεση του διεθνούς ρόλου του ευρώ δεν είναι στην εντολή μας. Αλλά τούτου λεχθέντος ο ρόλος του έχει μειωθεί σε κάποιες ε, διαστάσεις. Πιο συγκεκριμένα στην χρήση του ως αποθεματικό νόμισμα. Αλλά τούτου λεχθέντος ε, παραμένει το δεύτερο πιο χρησιμοποιούμενο νόμισμα στον κόσμο. Και εμείς ε, το βλέπουμε ως εξής ο διεθνός του ρόλος ε, κυρίως κρίνεται από τις δυνάμεις της αγοράς. Το ευρωσύστημα δεν εμποδίζει ούτε προωθεί τον ε, διεθνή ρόλο του ευρώ. Είμαι σίγουρος ότι αν και όσο θα προχωράμε προς την Ένωση Κεφαλαίου Αγορών ε, και την Τραπεζική Ένωση, θα ισχυροποιηθεί ο διεθνής ρόλος του ευρώ. Ο ρόλος του παγκοσμίω ε, λοιπόν σχετίζεται με την αποφασιστικότητα και την ικανότητα που έχουμε να κάνουμε μεταρρυθμίσει. Του τελευταίντος αναμένουμε και το τι θα προτείνει συγκεκριμένα η Κομισιόν και οπωσδήποτε ε, είμαστε στη διάθεση της Κομισιόν για συνεργασία. Σας ευχαριστώ. Αν θέλετε, έχετε χρόνο για άλλη μια ερώτηση. Όχι, Σβέν Γκίγκολτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ντράγκη, σε μια ομιλία σας σε μια ομιλία πριν από δέκα ημέρες ε, επευκαιρία τη επαιτίου τη κατάρρευση ε, τη ε, Λίμαν, ο προκάτοχό σα, ο κ. Τρισέ, είπε ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα παγκοσμίω αυτή τη στιγμή είναι τουλάχιστον τόσο ευάλωτο όσο ήταν πριν από 10 χρόνια. Και προειδοποίησε για τον υπερβολικό όγκο, την υπερβολική μόχλευση θα έλεγα, του χρηματοπιστωτικού συστήματο σε σχέση με την πραγματική οικονομία. Και μόλις ε, εσείς δικαιολογήσατε και ανακοινώσατε ότι θα συνεχίσετε να έχετε αυτήν την νομισματική πολιτική και τώρα όμως οι πολίτες στην Ευρώπη βλέπουν τις αρνητικές πτυχές αυτής της πολιτικής. Βεβαίως η νομισματική πολιτική είχε ένα σημαντικό ρόλο να παίξει στην Ευρωζώνη και ποτέ δεν ήμουν κάποιος από αυτούς και το Κοινοβούλιο. Άλλωστε κατά πλειοψηφία δεν άσκησε κριτική στην γενική σας θέση. Αλλά ακούγοντας ε, και τον προκάτοχό σας. Μήπως έχει φτάσει η στιγμή να δείτε τις αρνητικές ε, πτυχές ε, πιο πολύ. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξής. Συμφωνείτε με την παρατήρηση του προκατόχου σας. Και δεύτερον, εάν ναι, αυτή η υπερβολική μόχλευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε σχέση με την πραγματική οικονομία, εάν είναι όντως πρόβλημα, τι ε, αντλεί ως συμπέρασμα από αυτό η έκτη για την πολιτική της. Θα ήθελα καταρχήν, ε, επιτρέψτε μου να σχολιάσω κάπως αυτή την απάντηση, γιατί πρέπει να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ της, ε, του τραπεζικού συστήματος και του σκιωδούς τραπεζικού συστήματος. Να σας πω, στο κομμάτι του τραπεζικό δεν έχουμε κάποια πρόοδο. Αυτή τη στιγμή έχουν ε, κεφάλαιο CET1, ε, το οποίο είναι πραγματικά αρκετά υψηλότερο από αυτό που είχαν στο παρελθόν. Οπότε είναι πιο στεναρές σε επίπεδο ε, ρευστότητας, σε επίπεδο μόχλευσης. Οπότε δεν υπάρχει κανένας δείκτης ο οποίος δεν έχει προοδεύσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. και κανένα κομμάτι της διαχείρισης κινδύνου του τραπεζικού συστήματος δεν έχει μείνει αμετάβλητος από τότε που ξεκίνησε η κρίση. Οπότε, από αυτή την οπτική γωνία για τον τραπεζικό κλάδο, πρέπει να σου πω πως οι τράπεζες είναι πιο δυνατές από τον στο παρελθόν. Τώρα τι σημαίνει αυτό, πως μπορούμε να προλάβουμε την επόμενη κρίση. Βεβαίως και όχι. Αλλά καθήκον μα ήταν να τις δυναμώσουμε. Το άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με τον σκιώδη τραπεζικό κλάδο και τουλάχιστον ε, σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκεί έχουμε σημειώσει πρόοδο. Και να σας πω πως αυτός ο κλάδος έχει αυξηθεί πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Θα έλεγα 8% κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια και φέτο είναι η τελευταία χρονιά, η μόνη χρονιά που είχαμε μια σταθεροποίηση. Οπότε ο κλάδος της ε, ε, σκιώδης, ο σκιώδης τραπεζικός κλάδος έχει οντότητε μεγάλες, περίπλοκες, διασυνδεδεμένες και σε κάποιο βαθμό ε, έχουν και τραπεζικές δραστηριότητες ή δραστηριότητες που ομοιάζουν τις τραπεζικές δραστηριότητες με είναι λιγότερο ορατέ. Οπότε, πολλά έχουν γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να συνεχίσουν να γίνονται. Όμως, άλλες δικαιοδοσίες δεν ήταν τόσο δραστήριες και η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε άλλες δικαιοδοσίες είναι αρκετά μεγάλη έτσι ώστε εάν έχουν εκείνες κρίση, ναι, θα μεταφερθεί και σε εμά. Να σας πω πως όπως θα θυμηθούμε σε μια εκδήλωση για τα 10 χρόνια από την χρηματοπιστική κρίση της ΕΠΑ, οι εποπτικές αρχές είπαν έχουν μειωθεί σε κάποιο βαθμό οι εποπτικές τους αρμοδιότητες, γιατί σε άλλα μέρη του πλανήτη έχουν την, έχουμε την εντύπωση πως μειώνουν το κανονιστικό πλαίσιο. Είναι δηλαδή, ε, πηγαίνουν προς, σε μια, προς μια άλλη κατεύθυνση. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά επαναλαμβάνω, έχουμε έκθεση και στις υπόλοιπε γωνιές του πλανήτη. Τώρα για τη μόχλευση. Και εδώ θα κάνω μία διάκριση μεταξύ της Ευρώπης και των υπολείπων κρατών. Ε, το ιδιωτικό χρέος στην Ευρωζώνη έχει μειωθεί. Και η μόχλευση επίσης έχει μειωθεί αρκετά. Στο δημόσιο χρέος όχι, όχι. Εξακολουθεί να παραμένει υψηλό. Αλλά αυτό σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται και από άλλους παράγοντες. Εξακολουθούμε εμείς να παρακολουθούμε λοιπόν τον κίνδυνο για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα ε, στενά. Κοιτάμε όλες τις παραμέτρους και είδαμε ότι σε κάποιους κλάδους οικονομίας οι αποτιμήσεις είναι πιεσμένες, για παράδειγμα ακίνητα, επίσης χρέος υψηλής απόδοσης, εκεί οι αποτιμήσεις είναι πιεσμένες ε, στην ε, κατοικία και τα κίνητα εκεί σε κάποια κράτη και σε κάποιες περιοχές αυξάνονται οι τιμές. Η κτηματαγορά νομίζω σε όλη την Ευρωζώνη αυξάνει τις τιμές της και αναρωτηθήκαμε πώς να ανταποκριθούμε σε αυτό. Και πριν από πολλά χρόνια όταν κάναμε τον πρώτο σχεδιασμό αυτής της πολιτικής αποφασίσαμε πως δεν είναι σωστό να αλλάζουμε την νομισματική πολιτική για το επειδή υπάρχει κίνδυνος σταθερότητας χρηματοπιστωτικής. Όχι, θα πρέπει να έχουμε κάποια μακροπροληπτικά εργαλεία τα οποία θα πρέπει να λειτουργήσουν όχι μόνο μέσω της ΕΚΤ αλλά και μέσω των εθνικών αρμοδίων αρχών. Εμείς είτε μέσω του SRB είτε μέσω της ΕΚΤ ε, ε, εκδίδουμε προειδοποιήσεις Νομίζω το επόμενο βήμα είναι η αύξηση των μέτρων από την εργαλειοθήκη για τη μακροπροληπτική πολιτική για να καλύπτουμε και το σκιώδη τραπεζικό τομέα. Ο κύριος Βιέγκας παρακαλώ. I will talk in Θα μιλήσω πορτογαλικά. Παρακαλώ, να έχετε την καλοσύνη να φορέσετε ακουστικά σας. Ήθελα λοιπόν απλώς να θέσω μία ερώτηση. Αυτή αφορά την εμπλοκή της ΕΚΤ και τη δική σας εμπλοκή στην ομάδα των 30, Group of 30 όπως αποκαλείται. Αυτή η εμπλοκή σας επεκρίθη επανειλημμένα. Είναι μια ομάδα που συναθρίζει μεγάλες τράπεζες, μεγάλους χρηματοστικούς ομίλους και τράπεζες που τελούν υπό την εποπτεία της ΕΚΤ. Πρόσφατα έγινε μια έρευνα και το πόρισμα αυτής δείχνει ότι αυτή η συμμετοχή υπονομεύει την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και θέτει ένα αμφιβόλο την ανεξαρτησία της ως εποπτικό όργανο. Έχω μια απλή ερώτηση λοιπόν. Γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν ακολουθεί τις συστάσεις του διαμεσολαβητή της Ευρωπαϊκής Ένωσης του συνήγορου του πολίτη. Το ίδιο θέμα έχει τεθεί και για την ε, Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας. Υπάρχει μια ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι τα πρακτικά αυτών των συνεδριάσεων που πραγματοποιούνται και κλεισμένων των θερών να δημοσιοποιούνται. Είναι θέμα δημοσίου ελέγχου και λογοδοσίας. αυτό που αναφέρατε στην αρχή στην ομιλία σας. απάντηση. Ευχαριστώ, όπως γνωρίζετε, Υπήρχε μεγάλη ανταλλαγή αλληλογραφία και σημειώνουμε την απόφαση του Ευρωπαίου Διαμεσολογητή τη 3 η Ιουλίου 2018 για την εμπλοκή των μελών των φορέων ύψο αποφάσεω τη ΕΚΤ στην ομάδα των 30 καλωσορίζουμε προτάσει για περαιτέρω βελτίωση τη διαφανεία στην ΕΚΤ και το πλαισίο ορθή διακυβέρνηση. Η ΕΚΤ, κατά παρελθόν, έχει δώσει λεπτομερεί εξηγήσει στι θέσει τη όσον αφορά το θέμα αυτό. Καταρχά, στην επιστολή τη προ τον Ευρωπαίο Δημοσιονομητή του 31 Οκτωβρίου 2017 και μετά στην τεκμηριωμένη ε, γνωμοδότηση του Απριλίου 2018 είναι δημοσία διαθέσιμα τα έγγραφα αυτά στην ισοσελίδα μας. Σε αυτές τις απαντήσεις επίσης παρουσιάσαμε τα σημαντικά βήματα που έλαβε η ΕΚ τα τελευταία χρόνια ούτω ώστε να ενισχύσει τη διακυβέρνησή της. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα ανταποκριθεί στην απόφαση του Ευρωπαίου Δημοσιολογητή τις επόμενες ημέρες όπως πάντα έκανε κατά το παρελθόν και θα δημοσιοποιηθεί η απάντηση. Επίσης απαντήσαμε στις διάφορες γραπτές ερωτήσεις που λάβαμε από ευρωβουλευτές του τελευταίους ε, μήνες επί του θέματος αυτού. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ορίστε. Λυπάμαι που επιμένω αυτό που λέτε βασικά είναι ότι ο πρόεδρος Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα παραμείνει πλήρες μέλος της ομάδας των 30. Σωστά, σας κατάλαβα από την απάντησή σας αυτό εννοείτε. Απάντηση, δεν έχω τίποτα να προσθέσω σε αυτά που σας είπα. Θα ανταποκριθούμε, συμμορφωθούμε με την απόφαση του Ευρωπαίου Διαμοσολαβητή τις επόμενες ημέρες. Όπως κατά το παρελθόν η απάντηση θα δοθεί δημοσία. Σας ευχαριστώ. Μπερνάρ Μονού. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας. Για το ξέπλυμα χρήματος. Μας είπαν πως η Danske Bank στην Εστονία, στο παράρτημα εκεί, έχει κάνει 200 δις ξέπλυμα μεταξύ 2012 και 2015. Η κυρία Μπερές μίλησε για την IBLV. Ακόμα χειρότερα, ο διοικητή τη Λετωνική Κεντρική Τράπεζα που ανήκει και στο διοικητικό σας ε, ε, συμβούλιο, ζητούσε 100.000 ευρώ το μήνα για να κάνει υποπτία με τα μάτια κλειστά. Με συγχωρείτε. Τεκμήριο βέβαια. Εντάξει. Αλλά συγγνώμη, είναι ακόμα στη θέση του και δεν έχει καμία όρεξη να παραιτηθεί ο Πρωθυπουργό της Λετωνία, όταν γινόντουσαν αυτά, ο κύριος Ντομπρόφσκης, που δεν έχει έρθει εδώ ακόμα, δεν είχε καταλάβει τίποτα. Και είναι τώρα αντιπρόεδρο και ερμόδιο για την Ευρωζώνη. Πείτε μου, συγγνώμη, τι σημαίνει αυτό για την ελεύθερη κυκλοφορία στη ζώνη του ευρώ. Έτσι εμείς υποχρεώνουμε τα κράτη να ε, ε, εργάζονται σωστά. Εσείς, η ΕΚΤ λέτε, να είμαστε πιο ανοιχτοί, όλο και λιγότερο εθνικά σύνορα. Τέλη Σεπτεμβρίου, με τον κύριο Πρά, αυτό κάνατε ε, στη μεγάλη διάσκεψη ε, του ε, παγκοσμίου τραπεζικού λόμπινγκ. Πώς θα δώσουμε τη μάχη κατά του ξεπλήματος. Δεν μου κάνει εντύπωση που δεν λειτουργεί αυτή η μάχη, γιατί λέτε θα το αναλάβει κάθε κράτους μέλος και μετά σε ομόσπονδε επίπεδο κάποιου είδους ε, αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε ποιος θα κερδίσει. Οι παγκόσμιες εμβέλειες τραπεζα και, το, και, και ο σκιώδης τραπεζικός ε, κλάδος. Πείτε μου εσείς, τι θα κάνετε για το ξέπνα χρήματος μέσω ΕΚΤ χωρίς να ξεδοντιάσετε τα κράτη-μέλη. Πώς θα υποχρεώσετε να είναι ηθικά σωστοί οι συνάδελφοί σας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ. Λυπάμαι πως η θέση σας είναι λίγο ε, αντιφατική. Γιατί λέτε πως το σύστημα αυτή τη στιγμή είναι πολύ λίγο ικανοποιητικό, είναι καταστροφικό αλλά βασίζεται στο τι κάνουν το κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή. Για να το αλλάξουμε και για να το βελτιώσουμε, προτείνουμε περισσότερο συντονισμό και να έχουμε μία αρχή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε δεν μπορείτε να τα έχετε και τα δύο. Δεν μπορείτε να έχετε ένα σύστημα εθνικό το οποίο δεν συντονίζεται καθόλου, χωρίς να υπάρχει κάποια ομόσπονδη αρχή. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι τα λεγόμενά ήταν κάπως αντιφατικά. Να σας πω όμως το εξής και θα το επαναλάβω. Δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι για την επιβολή της νομοθεσίας, για την κατάχρηση του οικονομικού συστήματος έτσι ώστε να κάνει κανείς ε, νομιμοποίηση παράνομου χρήματος. Έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε. Εμείς πιέζουμε για μια ευρωπαϊκή αρχή. Έχουμε κάνει πάλι αυτό το σημείο εισόδου, μια πύλη, ένα πόρταλ στην ΕΚΤ που είναι ομόσπονδη αρχή και όχι εθνική αρχή. Γιατί είναι προφανές ότι το τρέχον σύστημα δεν λειτουργεί. Euh, Κύριε Πρόεδρε, δεν απαντάτε στην ερώτησή μου. Κύριε αφορά τον κύριο Ιμψεβικ. Και δεύτερον, δεν βλέπω καμία αντίφαση σε σχέση με τη διαχείριση και τον έλεγχο του ξεπλήμαχο βρώμικου χρήματο. Η τάπεζα τη Γαλλία στη Γαλλία το πραγματοποιούσε τέλεια πριν την ύπαρξη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Υπήρχαν έλεγχοι που διεξήγονται εξίσου και από το Υπουργείο Οικονομικών στη Γαλλία. Δεν υπήρχε κανένα τέτοιο πρόβλημα υπήρχε διαχείριση σε επίπεδο κράτους. Η θέση του κ. Ρίντσεβιτς είναι μια θέση που αφορά την εθνική δικαιοδοσία της χώρας του. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο από αυτό που ήδη έχει γίνει μέσω προσφυγή στο ε, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου. Το δικαστήριο απεφάνθη. Τώρα έχει διοριστεί κάποιος αναπληρωτής. Άρα έχει βελτιωθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Η κατάσταση δεν είναι αυτή που είναι επιθυμητή, δεν μας αρέσει. Αυτό όμως διότι ε, συνεχίζεται ε, η δικαστική υπόθεση στη χώρα του κυρίου Λίνσεβιτς. Το άλλο που το να πούμε ότι μια εθνική αρχή ή δύο ή τρεις εθνικές αρχές εκτελούν το καθήκον τους άριστα δεν σημαίνει ότι η βάση πρέπει να κινηθούμε βάσει κράτου μέλου, να διερωτηθούμε πώ το ξέπλυμα του χρήματο, το πιο αδύναμο τμήμα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, λειτουργεί, πώ έχει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Και εκεί ισχύει το επιχείρημα να έχουμε ένα συντονισμένο σύστημα ισχυρό, όπου γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών. Χωρί ανταλλαγή πληροφοριών δεν υπάρχει ούτε μία ελπή να είναι κανεί αποτελεσματικό για την αντιμετώπιση του ξεπλήματο βρωμικού χρήματο. Ευχαριστώ. Μάρκους Πρέτσελ. Κύριε Πρόεδρε, δέκα χρόνια μετά τη χρεοκοπία της Λίμαν, με το αποτέλεσμα του μηδενισμού των επιτοκίων, ε, ουσιαστικά έχει δύο μόνο εργαλεία η ΕΚΤ. Τα αναφέρατε το Asset Purchasing Program και δεύτερον το Forward Guidance, η κατεύθυνση που δίνει για το μέλλον. Εν τω μεταξύ ο ισολογισμός σας έχει διονγκωθεί, έχει φτάσει σε πάνω από 4,53 εκατομμύρια ευρώ, 41% δηλαδή του ΑΕΠ της Ευρωζώνης. Το πρώτο μου ερώτημα λοιπόν είναι, έχει πόρους και μέσα η ε, ΕΚΤ ε, για να μπορέσει να διαχειριστεί τον ισολογισμό της οποίος διωγγώθηκε τόσο πολύ. Δεύτερον, η Deutsche Bank ε, προσφάτως ε, έχει μία ενδιαφέρουσα ιστορία και εσείς μας είπατε βεβαίως ότι η κατάσταση των τραπεζών βελτιώθηκε σαφώς. Εν τω μεταξύ η Deutsche Bank εξακολουθεί να έχει ένα ποσοστό, μια πιθανότητα χρεοκοπίας εντός πενταετίας 7,7%, κάτι το οποίο είναι υψηλότερο από τον κίνδυνο που είχε η Ιταλική Unicredit Bank. Και φαίνεται ότι δεν βοήθησε η νομισματική πολιτική, τουλάχιστον τη συγκεκριμένη τράπεζα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, φαίνεται ότι έχει αγοράσει σχετικά μιλώντας ολίγα ιταλικά ομόλογα. Μήπως υπάρχει λοιπόν από δικιά σας πλευρά μια ανισορροπία μεταξύ των όσων κάνατε για την Ιταλία, την χώρα σας και για την Γερμανία όσον αφορά αυτό το μέσον. Είμαστε λοιπόν ενώπιον της συγχώνευσης της Deutsche Bank με την Commerzbank. Δύο πολύ αποδυναμωμένες τράπεζες θα συγχωνευτούν. Έχει καταποντιστεί η αξία του στο χρηματιστήριο έχουν φύγει από τον δίκτυ Eurostox 50 και από τον DAX αντιστοίχω η Deutsche Bank και η Commerzbank. Δεν μετράνε πλέον στους δείκτες σας. Ναι, καταλήξτε κάπου λέει ο πρόεδρος, έχετε δύο λεπτά. Ναι, με συγχωρείτε. Και μία τελευταία σύντομη ερώτηση. Είπατε πριν πως οποιοδήποτε περιορισμός ε, ρητός ή μη του Target 2 θα καταστρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια και της Γερμανίας να περιοριστεί τουλάχιστον στο 1 3 εκατομμύριο ευρώ θα ήταν επίσης ε, μοιραία. Πρέπει η Γερμανία να δεχτεί ότι ε, το target θα ξεπεράσει αυτό το ποσό. Η απάντηση στην τρίτη ερώτησή σας είναι ναι, θα ήταν μοιραία. Μια τέτοια παρέμβαση. Δεν έχει κάποιο νόημα να έχουμε νομισματική ένωση και να μπορώ να κάνω πληρωμές μέχρι ένα συγκεκριμένο ποσό και μετά να μην ξέρω τι να κάνω, ότι θα χρησιμοποιήσουμε άλλο νόμισμα. Δηλαδή δεν ξέρω πώς ε, θα εξελιχθούν αυτές οι ιδέες. Αυτή ήταν η τελευταία ερώτηση. Η πρώτη τελευταία ερώτηση. Δεν είστε ενήμερος. Λέτε ότι η ΕΚΤ αγόρασε ε, Ιταλικά δάνεια. Όχι. Δεν ισχύει. Απλά αγοράσαμε κρατικά και εταιρικά ομόλογα σε κάθε χώρα σύμφωνα με την σχετική κλίδα. Δεν υπάρχει προτιμησιακή μεταχείριση μιας χώρας. Ε, ασκούμε νομισματική πολιτική και θέμε σταθερότητα τιμών για ολόκληρη την Ευρωζώνη, όχι για μια χώρα. Η άλλη ερώτηση για την Deutsche Bank. Δεν ε, σχολιάζω συγκεκριμένες τράπεζες. Να πω ότι οι τράπεζες έχουν κάποια ιστορικά προβλήματα. Τα ιστορικά προβλήματα είναι τα προβλήματα τα οποία προήλθαν από τη μεγάλη ε, οικονομική κρίση και σε κάποια μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτά έχουν την μορφή των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Σε άλλα μέρη έχουν την μορφή των στοιχείων του λεγόμενου επίπεδου 2 και 3 ή τα οποία έχουν απαξιωθεί πολύ. Οπότε, και στις δύο περιπτώσεις ε, βεβαίως θα μπορέσει να προχωρήσει η Τραπεζική Ένωση αν αντιμετωπίσουμε αυτά τα ιστορικά προβλήματα. Δεν θα σχολιάσω τώρα συγκεκριμένες τράπεζες. Η πρώτη σας ερώτηση τώρα για τον ισολογισμό της ε, τράπεζας. Πράγματι έχει επεκταθεί πολύ. Ταυτόχρονα υπάρχουν ε, διατάξεις και προβλέψεις. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν κάποια κριτήρια επιλεξιμότητας ε, που σημαίνει ότι η ποιότητα των όσων έχουμε στον ισολογισμό μας είναι αρκετά υψηλή. Δεύτερον, έχουμε κάποια όρια εκθέσεων έκθεσης. Δεύτερον, έχουμε προβλέψεις ε, για επιτόκια, για συναλλαγματικές ε, ισοτιμίες, οπότε είμαστε αρκετά καλά προετοιμασμένοι. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζουμε. Η ΕΚΤ, όπως οι περισσότερες, αν όχι όλες οι κεντρικές τράπεζες, οπωσδήποτε αυτές ε, των μεγαλύτερων χωρών, τα στοιχεία ενεργητικού της δεν τα υπολογίζει με βάση την ε, τιμή της αγοράς αλλά με βάση την απόσβεση. Οπότε ε, οι αλλαγές ε, στα επιτόκια δεν τα επηρεάζουν άμεσα. Αυτά. Σας ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Κύριε Μακοσέλα, εδώ είμαι. Ένα Ιταλό πολίτη, ή Ευρωπαϊο πολίτη, όταν ακούει να λέει ο αντιπρόεδρο τη κυβερνήσεω τη Ιταλία για τον πρώτο προπολογισμό υπουργό οικονομικό θα, θα δημιουργήσει κάποιο έλλειμμα και μετά θα προσπαθήσουμε να το εξυπηρετήσουμε το χρέο αυτό τα επόμενα έτη. Ο πολίτη σκέφτεται λοιπόν και φαντάζεται ότι η Ευρώπη είναι εκείνη που δεν επιτρέπει να μπορέσει να δαπανίσει λόγω αυστηρών κανόνων, σαν κακή μητριά. Περιορίζει. Μπορούμε να πούμε λοιπόν, κατά την άποψή σας, αν το ένα, μπορεί να ξεπεράσει κανείς το όριο το 1,8%, αν είναι σκόπιμο η Ιταλία να ξεπεράσει αυτό το ανώτατο όριο, λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις 4 Μαρτίου το spread ανέβηκε κατά 130 ε, βαθμούς, αν θέλετε. Δηλαδή, από τη στιγμή όπου καλείται ο υπουργό της Οικονομίας να δημιουργήσει μεγαλύτερο χρέος, υπάρχει ένας κίνδυνος να επωνομευθούν τα οικονομικά της χώρας, οι λογαριασμοί της χώρας, προϋπολογισμός της χώρας. Απάντηση. Πρόεδρε, αν επιτρέπετε θα απαντήσω στα Ιταλικά, αν έχει την καλοσύνη. Κοιτάξτε, όπως είπα στη συνέντευξη τύπου της προηγούμενης εβδομάδας, πρέπει να σεβαστούμε τα στοιχεία, τα πραγματικά στοιχεία. Ποια είναι αυτά. Το νομοσχέδιο του προπολογισμού που κατετέθη και η συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Και τα δύο αυτά στοιχεία είναι σημαντικά και ευαίσθητα ζητήματα. Και σε αυτή τη φάση δεν θέλω να επισέλθω στο θέμα ή στις συζητήσεις που αφορούν κυβέρνηση μιας χώρας. Είπα την περασμένη φορά ότι τα λόγια έχουν δημιουργήσει ζημιές, διότι οικογένειες και επιχειρήσεις σήμερα πληρώνουν στις τράπεζες υψηλότερα ποσά από ό,τι πριν και υψηλότερους φόρους στις τράπεζες. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε και ότι οι τράπεζες στα νέα δάνεια από τον Απρίλιο και μετά, ακολουθώντας τη μείωση ε, των, της αξίας των αξιογράφων, οι τράπεζες αύξησαν τα επιτόκια περίπου κατά 20% κυρίως όσον αφορά τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για μεγάλες επιχειρήσεις που εκδίδουν ε, ομόλογα είναι χαμηλότερο το κόστος. Νομίζω 64 βασικά ε, βασικού πόντου όσον αφορά τι εκδόσει ομολόγων σε σύγκριση με τι μεγάλε επιχειρήσει. Το άλλο σημαντικό σημείο δεν είναι μόνο ότι αυξήθηκαν τα επιτόκια όσον αφορά τα δάνεια των τραπεζών, αλλά έγιναν πιο απαιτητικέ συνθήκε σχετικά με τι εγγυήσει και τι ρήτρε που υπάρχουν στα διάφορα, στις που συνάπτονται. Σε άλλες χώρες, οι επιχειρήσεις σε άλλες χώρες εξακολουθούν να πληρώνουν επιτόκια ως πριν, ίσως και πιο χαμηλά. Όσον αφορά τις οικογένειες, εκεί που είδαμε μία αύξηση των επιτοκίων, ε, επιτοκίων για τις οικογένειες, είναι για το καταναλωτικό δάνειο, για μικροδάνεια για οικογένειες. Και το πιστοτικό δάνειο, εκεί είδα μια αύξηση περίπου 20 σημείων, αν θέλετε, λίγο παραπάνω. Όσον αφορά βέβαια τα στεγαστικά δάνεια, οι εξελίξεις είναι πιο αργές, οι ευξήσεις είναι πιο αργές. Ορίστε. Αυτή η κατάσταση εξαρτάται από τα λόγια που ακούστηκαν, τα λαθασμένα λόγια. Και ίσως που δεν παρακολουθήθηκαν επαρκώς και ποιες θα ήταν οι συνέπειες, σωστά. Και, και δεν εξετάστηκαν τα στοιχεία. Απάντηση. Δεν πρέπει να ξεπεράσουμε τα όρια των εξηγήσεων. Αυτό που συνέβη στην Ιταλία δεν συνέβη αλλού στην Ευρωζώνη, συνέβη μόνο στην Ιταλία. Σας ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Λουίτζι Μόργαν ο επόμενος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για την παρουσία σας εδώ στο Κοινοβούλιο, σε αυτή τη συνάντηση. Τακτικές συναντήσεις είναι που θεωρώ ότι είναι πολύ καλό αυτό, ούτως ώστε η ΕΚ να μας δείχνει σε εμά το Κοινοβούλιο πώς λειτουργεί, αλλά και στο ευρύτερο κοινό, προφανώς στα πλαίσια της ανεξαρτησίας των δύο θεσμικών οργάνων Ευρωκοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Λοιπόν, λοιπόν πάνω σε αυτά που υπόθηκαν και λαμβάνοντας υπόψη αυτά που τα εισαγωγικά και το διάλογο με τους ε, προλαλήσαντες συναδέλφους, θα ήθελα να υποβάλω κάποιες ερωτήσεις που ίσως να θεωρούν κάπως παράδοξες. Σε αυτές τις συναντήσεις μας, τι θέλω να πω, η συζήτηση λοιπόν στι συναντήσεις μας, η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι αυτή ανθρώπων που γνωρίζουν την οικονομική πολιτική και κυρίως την νομισματική πολιτική ίσως δεν υπογραμμίστηκε αρκετά, αλλά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και εσείς πιο συγκεκριμένα ε, εξασφαλίσατε ότι θα, στην κρίση θα, θα προστατευτούμε στην Ευρωζώνη και στην Ευρώπη τις συνέπειες της κρίσης. Αντίθετα γνωρίζουμε ότι κάποιοι εθνικοί ηγέτες ε, ακολούθησαν δρόμο πολύ εθνικό και όχι ευρωπαϊκό όπως για τη, που δεν γίνει συζήτηση για τις καταθέσεις και για την αντικυκλική προσέγγιση των κρίσεων, για τη διαχείριση των κρίσεων και μετά την κρίση. Έχουμε σε λοιπόν. Βλέποντας τα τελευταία έτη, πώς θα μπορούσατε να συνοψίσετε το πώς κινήθηκε η ΕΚΤ, πώς θα το εξηγούσατε στους πολίτες που δεν συμμετέχουν στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, αλλά ζουν καθημερινά οι πολίτες, τις συνέπειε τη εργασία που γίνεται εκεί και των αποφάσεων που λαμβάνονται. Αν φανταστούμε ότι μιλάμε με τους πολίτες, τι θα υπογραμμίζατε όσον αφορά την κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας όπως είναι σήμερα και οι δυνατόν ποιοι είναι οι κίνδυνοι που διαβλέπετε στον ορίζοντα. Όχι διότι τους αναφέρατε αλλά ποιε συνέπειε θα μπορούσαν να υπάρχουν στον αφορά την νομισματική πολιτική. Γιατί το λέω αυτό, διότι όλο και περισσότερο, ίσω γιατί πλησιάζει το τέλος της ευρωπαϊκής Πενταετία που μας αφορά, υπάρχει και το αίτημα από πολλού ανθρώπους και από πολλού συμπολίτε μας να προσπαθήσουν να καταλάβουν αν δυνατόν να έχουμε μια πιο ανθυρή οικονομία, βλέποντα και ποιο είναι και το διεθνέ πλαίσιο που κινείται και εάν ήταν δυνατό να υπάρχει ένα καλύτερο μέλλον για την Ευρώπη. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Απάντηση. Μπορώ να απαντήσω Ιταλικά. Θα χρησιμοποιήσω και Ιταλικά και Αγγλικά. Λοιπόν, τα μέτρα νοσομητικής πολιτικής είχαν σημαντικό αντίκτυπο όσον αφορά την οικονομία της Ευρωζώνης και αυτό που εκτιμά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι τα τελευταία τέσσερα χρόνια, 2016 μέχρι το 2020, συμβάλλουν σε μεγαλύτερη ανάπτυξη. Το είπα και στο εισαγωγικό μου παρέμβαση, κατά 1,9% αύξηση και ένα πληθωρισμό σε ανάλογο επίπεδο. Εν γέννη όμως, η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ θα έλεγα ήταν θεμελιώδου σημασία στα χρόνια που δεν υπήρχαν άλλες πολιτικές για να μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση του ευρώ από το 2012 και μετά μέχρι τα μέτρα του ε, QE, της ε, ποσοτικής χαλάρωσης, των προσανατολισμών για τα επιτόκια και για την προσπάθεια ε, επανεπενδύσεων στα αξιόγραφα που εξέπνεαν. Ο ρόλος της ΕΚΤ υπήρξε. Εγώ είμαι παρατηρητής που συμμετέχει σε όλα αυτά βέβαια. Αυτή η κρίση θα έπρεπε να επιβεβαιωθεί, θα έλεγα, απαλού αλλού. Βλέποντας και λίγο γύρω τι γίνεται και τι λένε οι άλλοι πολίτες της ε, Ευρωζώνης. Ευχαριστώ. Ο Brian Hayes. Ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να σας καλωσορίσω για μια φορά ακόμα στην Επιτροπή μας. Ξέρω πως ο Μάρκος Φάρμπερ σας ρώτησε τι θα γίνει με το hard Brexit, αλλά θέλω εγώ να ε, πω δύο κουβέντες παραπάνω. Η Κριστίν Λιαγκάρτ πρόσφατα είπε πως ένα Brexit χωρίς συμφωνία θα έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις, όχι μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και για την Ευρωζώνη. Συμφωνείτε? Εγώ κατανοώ απόλυτα πως εσείς δεν αποτελείτε τμήμα της διαπραγματευτικής ε, ομάδες. Επαναλαμβάνω την παρατήρησή μου. Δραματικές και δύσκολες συνέπειες προβλέπει η Κριστίν Λιαγκάρτ σε περίπτωση σκληρού Brexit, όχι μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και την Ευρωζώνη. Παρακαλώ, σχολιάστε. Και δεύτερον, δεν είστε κομμάτι τη διαπραγματευτική ομάδα και συνεργάζεστε σε κάποιο βαθμό στην ομάδα εργασία με την Τράπεζα τη Αγγλία. Εσεί βλέπετε να υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη, κυρίω το δικό μου, η Ιρλανδία, που θα επηρεαστούν δυσανάλογα από ένα σκληρό Brexit και όπως είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε έχουμε πολύ υψηλό δημόσιο χρέος σε τη χώρα μου και σε όλη την Ευρωζώνη πώς θα επηρεαστούν. Και ρωτώ το εξή. Αν μια χώρα επηρεαστεί άσχημα, για παράδειγμα όπως η δική μου ή άλλες, τι θα πρέπει να κάνει η Ευρωζώνη ως μπλοκ για να διευκολύνει τις πιέσεις ε, που θα έχουν ε, οι επιπτώσεις του σκληρού Brexit. Και δεύτερον, πώς θα συμβουλεύσετε τις εθνικές αρμόδιες αρχές και τις δημόσιες αρχές στα κράτη-μέλη αυτά τα οποία έχουν μεγαλύτερη έκθεση στο σκληρό Brexit για το πώς μπορούν να δημιουργήσουν ε, ένα περιθώριο, ε, μια λωρίδα απομόνωσης, ένα μαξιλαράκι. Τι συμβουλή θα δώσει η ΕΚΤ η οποία αυτή τη στιγμή διευθύνει την νομισματική επιλογή, ε, πολιτική με στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό. Γιατί το νόμισμά μας είναι το ευρώ και ανήκει στα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Και είναι και γερμανικό και ιρλανδικό και γαλλικό νόμισμα. Υπάρχουν όμως συνθήκες σύμφωνα με τις οποίες δυσανάλογα κράτη-μέλη επηρεάζονται από το πολύ σκληρό Brexit. Και νομίζω είναι σημαντικό για τους πολίτες της χώρας μου, για παράδειγμα, να ακούσουν τι πιστεύετε εσείς θα είναι η σωστή απόκριση σε μια ενδεχομένως τέτοια περίπτωση όπου θα ε, κλείσει η υπόθεση με σκληρό Brexit. Ευχαριστώ πολύ. Σε κάποιο βαθμό κάνετε πολύ σωστά που ρωτάτε ε, αυτή την ερώτηση, αλλά είναι πολύ νωρίς για να σας δώσω μια πλήρη και ικανοποιητική απάντηση για τις επιπτώσεις. Όταν είπα προηγουμένως πως οι επιπτώσεις μέσω του εμπορίου και σε μεγάλο βαθμό και των ε, χρηματοπιστωτικών διάβλων δεν μοιάζουν να είναι υπερβολικά υψηλές με τη μία εξαίρεση που ανέφερα, μιλούσα για ολόκληρη την Ευρωζώνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν μεμονωμένες χώρες οι οποίες δεν έχουν σημαντική έκθεση στο σκληρό Brexit. Μια περίπτωση είναι η Ιρλανδία, ίσως είσαστε και η περίπτωση είναι πολύ δύσκολο να προβλέψουμε τι θα γίνει, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Όμως, θα σας αφήσει μόνος η υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση να το αντιμετωπίσετε. Μου φαίνεται απίθανο, δεδομένου το ότι οι αξίες μας συμπεριλαμβάνουν και την αλληλεγγύη. Νομίζω ότι αυτή είναι ξεκάθαρα προσωπική άποψη. Δεν έχει συζητηθεί κάτι αντίστοιχο. Θεωρούμε πως είναι απίθανο αυτό το σενάριο, αλλά αν εμείς να κάνουμε κάποιες σκέψεις έτσι για τα απίθανα γεγονότα, ναι, θα κατέληγα σε αυτό το συμπέρασμα. Μπράιαν, ξέρεις και εσύ πως επηρεαστεί δυσανάλογα η Ιρλανδία επίσης αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ε, διαπραγματευτεί και ένα λειτουργικό backstop. Ε, κάνουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις ακριβώς γιατί σας στηρίζουμε Ιρλανδία στο θέμα αυτό του backstop ως προϋπόθεση της λύσης δηλαδή για τα σύνορα μεταξύ Βορείου Ιρλανδίας και Ήρε. Καλώς ήρθατε κύριε Ντράγκη. Θα ήθελα και εγώ να θεωρώ πως η ΕΚΤ παρακολουθεί τις, εξετάσεις, τις εξελίξεις και μάλιστα τις καθορίζει. Αλλά έχετε μείνει πίσω στο θέμα της ε, βιώσιμης ε, χρηματοδότησης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε μια έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας η οποία λέει ότι θέλουμε ένα υποχρεωτικό πλαίσιο δέουσας επιμέλειας το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να ελέγχουν ε, και να προλαμβάνουν οι επενδυτές ε, τέτοιες, ε, τέτοια ανοίγματα, κάτι το οποίο σημαίνει βεβαίως ε, και επενδυτικά και συνταξιδοτικά ταμεία και θα μπορούσε να περιλαμβάνει και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορείτε να επαναλάβετε την ερώτησή σας γιατί κάποια μου ξέφυγαν. Η βιώσιμη ε, χρηματοοικονομική γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι και επενδυτής ε, μέσω της ε, πολιτικής της και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει οι επενδυτές ε, να λάβουν υπόψη τους παράγοντες αυτούς της βιώσιμης χρηματοοικονομικής και να φροντίσουν να υπάρξει μια αντιμετώπιση αυτών των παραγόντων και υπάρχει και ένα ενδιαφέρον, μια ενδιαφέρουσα εργασία από τον κύριο Σουμαχέρο ο οποίος ε, λέει με τίτλο «Πρασίνισμα της νομισματικής πολιτικής» και λέει ότι το ευρωσύστημα θα μπορούσε να στηρίξει τους κλιματικούς στόχους μέσω ενός πρασινίσματος της νομισματικής πολιτικής και λέει ότι αυτό μπορεί να γίνει χωρίς να διαταραχτεί η ομαλή λειτουργία της νομισματικής πολιτικής για να μην ε, υπάρχει και πρόβλημα με τον στόχο της ε, ε, του στόχου της σταθερότητας των τιμών. Το ερώτημα είναι λοιπόν εάν είναι διατεθειμένοι να περάσουν τον Ρουβίκονα. Λοιπόν, ακούσατε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι υπέρ ενός τέτοιου υποχρεωτικού πλαισίου. Είναι λοιπόν έτοιμη η ΕΚΤ να κάνει το ίδιο για να είναι μπροστά από τις εξελίξεις. Να πω ότι ε, οτιδήποτε βεβαίω ε, θα πω δεν επηρεάζει τον κύριο στόχο μα που είναι η σταθερότητα των τιμών. του λεχθέντος η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υποστηρίζει τους γενικού στόχου ε, της Ένωσης ε, και μεταξύ αυτών το άρθρο 3 τη συνθήκη, περιλαμβάνει την φόρα ανάπτυξη της Ευρώπη και ένα υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος. Οπότε αναγνωρίζουμε αυτή την πρόκληση που θέτει η κλιματική αλλαγή και την σημασία της αντιμετώπισης της. Οπότε στηρίζουμε την δουλειά που γίνεται σε διάφορα διεθνή φόρα και προσφάτως ενταχθήκαμε στο δίκτυο πρασινίσματος του χρηματοπιστωτικού συστήματος, στο οποίο συναντώνται κεντρικές τράπεζες και εποπτικές αρχές για να απτύξουν κάποιες κοινέ μακροπροληπτικές αρχές για ζητήματα που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον. Τώρα έρχομαι στο πρόγραμμα των εταιρικών ομολόγων. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας ε, του προγράμματος αγορών ε, των εταιρικό κλάδο δεν κάνουν αρνητικές ή θετικές ε, διακρίσεις ανάλογα με την οικονομική δραστηριότητα των εταιριών. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος στόχος μας είναι η νομισματική πολιτική που λαμβάνει υπόψη ε, τον χρηματοπιστωτικό κίνδυνο και την διαχείριση. Όταν όμως φτάνουμε στην, ε, στις δράσεις τις οποίες κάνουμε μέσω του προγράμματος αγοράς εταιρικών ομολόγων και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχω ξαναπεί στο παρελθόν η ΕΚΤ ε, έχει αγοράσει ένα σημαντικό αριθμό πράσινων ομολόγων και μάλιστα το ποσοστό πράσινων ομολόγων ως ε, ποσοστό του συνολικού χαρτοφυλακίου είναι το ίδιο με το ποσοστό που έχουν εντός των επιλέξιμων ομολόγων, εντός του πλαισίου επιλέξιμων ομολόγων. Το ποσό τώρα το ίδιο Δεν το έχω πρόχειρο, θα σας πω σε λίγο για να μην, ε, να μην πω κάτι λάθος. Είναι σημαντικό όμως. Ταυτόχρονα η ΕΚΤ έχει αγοράσει τα ομόλογα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που επίσης ε, ε, και αυτή αγοράζει πάρα πολλά πράσινα ομόλογα. Οπότε, εντός των ορίων της εντολής μας, οπωσδήποτε το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Σας ευχαριστώ, Λούντε Κνίντερμαγερ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που είστε εδώ και να σας ευχαριστήσω και πάλι. Εγώ θα αναφερθώ σε κάτι το οποίο συζητήσαμε πριν, το θέμα της επικοινωνίας και των κατευθύνσεων για το μέλλον. Έχω δύο ερωτήσεις. Πρώτον, προφανώς οι κατευθύνσεις αυτές για το μέλλον, ειδικά όσον αφορά τα επιτόκια, σας βοηθούν να μεταδώσετε το μήνυμα της νομισματικής πολιτικής και να επηρεάσετε σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου. Η κατεύθυνση αυτή λοιπόν για τα επιτόκια μπορεί όπως είπα, να σας βοηθήσει να μεταδώσετε το μήνυμά σας και να επηρεάσετε τα πράγματα μακροπρόθεσμα. Ταυτόχρονα μπορεί κάποιος να πει ότι εάν είναι πολύ εκτεταμένη αυτή η κατεύθυνση και το μεταξύ αλλάξουν οι συνθήκες, μπορεί να βρεθείτε σε μια κατάσταση όπου δεν θα είναι ιδανική η αντίδραση και αν αντιδράσει η Κεντρική Τράπεζα πολύ αργά, το κόστος προσαρμογή είναι υψηλότερο. Οπότε το πρώτο ερώτημα είναι πώς βλέπετε την ισορροπία μεταξύ αυτών των δύο στόχων. Το δεύτερο είναι ότι πώς βλέπετε να διαμορφώνεται αυτή η κατεύθυνση στο μέλλον. Αφενός μπορεί κανείς να πει ότι πρόκειται για μια ε, δέσμευση, αλλά εάν είναι κάτι τέτοιο, τότε το θέμα τίθεται το θέμα της βέλτιστης νομισματικής πολιτικής. Απ' την άλλη, αν είναι μια δέσμευση υπό όρους, τότε και εξαρτάται από τις μελλοντικέ εξελίξεις της οικονομίας, τότε θα μπορούσε κανείς να πει ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια στις προβλέψεις του ε, πληθωρισμού θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Πώς το βλέπετε. Για τους προσανατολισμούς, ε, τα πράγματα πήγαν αρκετά καλά. Κάθε φορά που εκφράζουμε τέτοιους προσανατολισμούς, υπάρχει μια προσδοκία που μπορεί να συνδεθεί με κάποια ανάληψη υποχρέωση. Να σας πω τι είπα ακριβώς αυτό το λεξί. Τα επιτόκια αναμένεται να παραμείνουν σε παρόντα επίπεδα και βαθμίζεται στις ε, παρούσες πληροφορίες μέχρι εμπεριέχεται βαθμός ε, επιλεξιμότητας ελιγμών, οπότε μπορούν να καλυφθούν και περιστάσεις απρόβλεπτες που ίσως προκύψουν. Τον, τον Ιούνιο του 2018 είπαμε ότι αναμένονται τα επιτόκια να παραμείνουν στα παρόντα επίπεδα τουλάχιστον και μέχρι το θέος του 2019 εν πάση περιπτώσει στο βαθμό που είναι αναγκαίο και εν πάση περιπτώσει όσο αυτό είναι απαραίτητο για να εξασφαλίζεται ότι η εξέλιξη του πληθωρισμού ευθυγραμμίζεται με τις τρέχουσες προσδοκίες ενός, μιας βιώσιμης προσαρμογής. Δηλαδή, κατευθύνει στις προσδοκίες για τα επιτόκια και πάνω σε αυτό βασίζεται και η προβολή για την εξέλιξη του πληθωρισμού. Τον Ιούλιο κάναμε προβλέψεις και έχει δύο τμήματα αυτό που είπαμε. Πρώτα απ' όλα έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα, ημερολόγιο. Δίνουμε προσανατολισμούς με ημερολόγιο μέσα από το καλοκαίρι, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2019. Και εκεί είναι που προβλέπουμε ότι θα υπάρχουν συνθήκες που ίσως να απαιτούν μια πρώτη αύξηση επιτοκίων. Και μετά εξαρτάται και από το κράτος. Δηλαδή τα επιτόκια θα παραμείνουν αμετάβλητα. Είναι η προσδοκία μας, εν πάση περιπτώσει, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για να εξασφαλίσουμε συνεχή βιώσιμη σύγκληση του πληθωρισμού σε επίπεδα που είναι κάτω από το ή πολύ κοντά στο 2%. Υπάρχουν διάφορα μονοπάτια τα οποία θα μπορούσαν να είναι επαρκή για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε διάφορες περιπτώσεις. Μετά μπορεί να πει κανείς ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά την πρόβλεψη του πληθωρισμού ε, μπορεί να δώσει τέτοια αποτελέσματα. Δηλαδή η πρόβλεψη του πληθωρισμού και η διαφάνεια αντιστοιχούν περίπου. Συμφωνώ απόλυτα με την προσέγγιση σας. Διότι ε, θα πρέπει να υπάρχουν δεσμεύσει για τη μελλοντική πορεία τη νοσηλευτική πολιτική. Και είναι κάτι που λειτουργήσε τα τελευταία χρόνια, ίσω όχι στο μέλλον και ίσω θα μπορούσε να υπονεμεύσει την αξιοπιστία. Είμαι πιο ικανοποιημένο με αυτή την προσέγγιση. Εγώ θα έλεγα ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια ε, στην πρόβλεψη μπορούσε να πετύχει το ίδιο. Απάντηση. Κοιτάξτε, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Αν δούμε τι έγινε κατά το παρελθόν, ίσως να εξαρτάται από την αξιοπιστία της κεντρικής τράπεζας. Αν η κεντρική τράπεζα γίνει αντιληπτή ότι είναι 100% αξιόπιστη, εν τη ενία ότι αρκεί να ανακοινώσει ένα στόχο η τράπεζα και τότε ο κόσμος θα καταλάβει ότι αυτός ο στόχος είναι σίγουρα εφικτός 100% τότε είναι το ίδιο. Υπάρχει μια κάποια διαμόρφωση, κάποια αλλαγή εκεί, διακύμανση εκεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ντράκη. Πρώτη μου ερώτηση έχει να κάνει με τα διδάγματα από την περασμένη δεκαετία για το σύστημα της ΕΚΤ. Και πιο συγκεκριμένα σας ρωτώ, φτάσαμε στο στο βαθμό ε, κεντρικοποίησης του συστήματος, γιατί οι αρμοδιότητες και για τον ΕΛΑ και για το PSPP, για τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες, χρήζουν αναθεώρησης. Επίσης, για το Target 2, εδώ θα μπορούσαμε να μειώσουμε λόγω του συστήματος που είναι πολύ πιο κεντρικοποιημένο. Τι θα κάνετε εσείς για τα θέματα αυτά, γιατί βεβαίως χρειάζονται κάποιες νομοθετικές αλλαγές. Δεύτερον, είχατε, δώσατε μια εξαιρετική έκθεση της ΕΚΤ και λυπάμαι που εσείς το έχετε ήδη απαντήσει, αλλά για τις προτάσεις της Κομισιόν για, τις, για τα SBs και την εισαγωγή αυτών, ε, θέλω να πω πως υπάρχει μια διαφορά μεταξύ της δικής σας πρότασης ε, και τις πρώτες κομισιόν και για το αν ε, τα μικρά παραρτήματα των τραπεζών, τα junior, η ε, junior tranche θα πρέπει να θεωρείται ως μη επικίνδυνη. Γιατί έτσι θα μπορούσαμε να έχουμε ένα πολύ ασφαλές κομμάτι το οποίο θα το προσθέτουμε στο senior trans. Εκεί έχετε πάρει κάποια απόφαση. Thank you. On, <clears throat> On your first question, um, Είναι αλήθεια πως στο παρελθόν μίλησα στην κεντρικοποίηση του μηχανισμού στήριξη του ELA. Προτιμώ όμως άλλη τερμο, ε, ορολογία τώρα που είναι διατάξεις περί ευρωπαϊκών καθεκόντων του ELA. Γιατί το σημαντικό για τον ELA με το μηχανισμό στήριξη είναι ο τρόπο που θα λαμβάνονται οι αποφάσει σε κεντρικό επίπεδο, ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι εθνικό. Αυτή η ορολογία δίνει κάποιες αναλογίες, για παράδειγμα, για το πώς εμείς κάνουμε κάποιες επιχειρήσεις νομισματικής πολιτικής, όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται κεντρικά, αλλά η προσφορά ρευστότητας γίνεται μέσω των εθνικών κεντρικών τραπεζών. Παρ' όλα αυτά η έννοια αυτή ακόμα είναι ανοιχτή προς συζήτηση. Αυτή τη στιγμή δεν θα σχολίαζα το θέμα της κατανομής κινδύνου. Αυτή τη στιγμή η προσφορά του μηχανισμού στήριξης ELA και οποιαδήποτε συνδεδεμένα κόστη και κίνδυνοι αναλαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο και οι εθνικές ε, κεντρικές τράπεζες απηχούν τα όσα έχουμε στην νομοθεσία. Οπότε ο ρόλο της ΕΚΤ περιορίζεται στην προσφορά του ELA που δεν θα πρέπει να έρχεται σε αντίφαση με τους στόχους μας στην νομισματική πολιτική. Όπως έχω πει στο παρελθόν θα μπορούσαμε να έχουμε μια μετακίνηση, μετάθεση αρμοδιοτήτων για την προσφορά του ELA ε, ε από τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αλλά ξέρετε πως γι' αυτό υπάρχει μια σειρά νομικών, πολιτικών και θεσμικών εμποδίων που θα έπρεπε να ξεπεράσουμε. Για τη δεύτερη ερώτηση που κάνατε. Να κάνω καταρχήν μία γενική. Ε, λοιπόν, το να έχει κανείς ένα ασφαλές ε, ε, στοιχείο ενεργητικού είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ουσιαστικά για τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και η αποτελεσματικότητα της διατραπεζικής διαμεσολάβησης είναι κομβική. Έχουμε τα ίσμπις καταρχήν Τα sovereign bonds λοιπόν που επιτρέπουν τη διαφοροποίηση και που επιτρέπουν να κάνουμε μια ε, κατάτμιση ε, του ε, πουλ των ε, στοιχείων ενεργητικού. Αυτό που είπατε λοιπόν εσείς βρίσκεται στην έκθεση ε, της ΕΚΤ και όλα τα τμήματα από τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες για λόγους ρευστότητας θα αντιμετωπίζονται το ίδιο, αλλά μπορεί να δημιουργηθούν κάποια προληπτικά θέματα, γιατί βέβαια κάποια από αυτά τα τμήματα μπορεί να θεωρούνται πιο επικίνδυνα από άλλα. Η δική μου άποψη είναι πως όλες αυτές οι προσπάθειες, γιατί βέβαια κανείς μπορεί να αξιολογεί και άλλες προτάσεις, για παράδειγμα λάβαμε προτάσεις ε, και πριν από αυτές για τα sovereign bonds, τα εθνικά ομόλογα δηλαδή, αλλά ακολουθούσαν μια πορεία πολύ πειραματική, γιατί θα ε, τακτική, γιατί έχουμε ένα βασικό πρόβλημα ε, στις χώρες μας. Είχαμε τα κρατικά ομόλογα, τα οποία παλιά θεωρείται ε, ασφαλές στοιχείο ενεργητικού και πλέον όχι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρούμε κάποιο άλλο ασφαλές στοιχείο ενεργητικού του ίδιου εύρους και της ίδιας εμβέλειας για να καλύψει τον ίδιο χώρο με προηγουμένους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στην αρχική σας παρέμβαση μιλήσατε για την οικονομία του ευρώ η οποία βρίσκεται σε προφανή αύξηση με κάποιες αβεβαιότητες βεβαίως στον ορίζοντα και είπατε επίσης η πιο μεγάλη αμφιβολία έχει να κάνει με τους γεωπολιτικούς κινδύνους. Σε αυτούς τους γεωπολιτικούς κινδύνους έχουμε τις, ε, τους πειρασμούς για προστατευτισμό από τη ΣΥΠΑ, αλλά βλέπουμε επίσης και τις επιπτώσεις της νομισματικής πολιτικής ε, του Federal Reserve, της Αμερικανικής ε, Τράπεζας, λόγω των μεγάλων δημοσιονομικών ελλημάτων στη ΣΥΠΑ και δημιούργησε αυτό στις αναδυόμενες οικονομίες, Βραζιλία, Αργεντινή κτλ. μεγάλες αναταράξεις, Τουρκία, πέρσι το καλοκαίρι. Φέτος μάλλον το καλοκαίρι. Και μια και είμαι ένας από τους τελευταίους που παίρνουν το λόγο, και επειδή τις ερωτήσεις που είχα σημειώσει εγώ τις έχουν κάνει άλλοι συνάδελφοι, θα ήθελα να μου πείτε το εξής. Αυτή η γεωπολιτική κίνδυνη τους οποίους βλέπουν να ε, υπάρχουν στη Βραζιλία, στην Τουρκία, στην Αργεντινή και που μπορεί να επηρεάσουν και την Ευρωζώνη, όπως επίσης ο κίνδυνος για προστατευτισμό μπορεί να ανατρέψουν ε, τα δικά μας ε, θέματα, γιατί έχουμε μια ανατροπή της νομισματικής πολιτικής αυτή τη στιγμή που γίνεται όλο και πιο συχτή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Thank you. Now let's go. Um, δούμε τον κατάλογο αυτών των πιθανών κινδύνων. Ο πρώτος είναι ο κίνδυνο από κάποιες αναψώμενες χώρες. Αναφέρατε την ε, Τουρκία και την Αργεντινή, κάποιες ανερχόμενες αγορέ. Ε, συνολικά φαίνεται ότι δεν έχουν μεγάλη σημασία για τις προοπτικές ανάπτυξης της Ευρωζώνης. Όμως μπορεί να υπάρχουν μεμονωμένα ιδρύματα που να είναι ιδιαίτερως εκτεθειμένα στον πιστοτικό κίνδυνο αυτών των χωρών. Αλλά σε γενικές γραμμές αυτό το οποίο βλέπουμε είναι, εντάξει βεβαίως μπορεί η διάδοση να αποτελέσει πρόβλημα, αλλά η διάδοση από αυτές τις δύο-τρεις χώρες σε άλλες χώρες να ακολουθεί μια συγκεκριμένη πορεία. Οι χώρες οι οποίες επηρεάζονται είναι επίσης οι χώρες οι οποίες έχουν πολύ ασθενή βασικά στοιχεία, δηλαδή υψηλό έλλειμμα ίσως γεωτροξών ε, συναλλαγών, υψηλό έλλειμμα του προπολογισμού, υψηλό πληθωρισμό κάποιες και βλέπουμε ότι η διάδοση αυτή είναι περιορισμένη σε άλλες ε, ανερχόμενες ε, αγορές. Οπότε συνολικά δεν νομίζω ότι μιλάμε για σημαντικό κίνδυνο για το σύνολο της Ευρωζώνης. Βεβαίως, διαφορετικό είναι το συμπέρασμα όταν μιλάμε για την απειλή του προστατευτισμού. Εκεί η τελική αξιολόγηση θα είναι δυνατή όταν θα γνωρίζουμε ποιος είναι ο βαθμός της κλιμάκωσης των πολιτικών τους επόμενους μήνες. Και αυτό έχει δύο διαστάσεις. Η μία είναι θέμα εμπιστοσύνη γιατί τα μέτρα προστατευτισμού είναι περίπλοκα και είναι δύσκολο να αντιληφθούμε το ποιος είναι ο αντίκτυπος ε, στο ΑΕΠ ε, σε διάφορα σημεία του κόσμου συνολικά είναι αρνητικός. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο τα όσα έχουν ανακοινωθεί και εφαρμοστεί. Και ο αντίκτυπός τους αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ μεγάλος, αλλά έχουν ανακοινωθεί και άλλα μέτρα που δεν έχουν ακόμα εφαρμοστεί. Και ε, πρέπει να δούμε ποια θα είναι και η αντίδραση άλλων χωρών. Και όλα αυτά έχουν και ίσως ήδη έχουν επηρεάσει αρνητικά την εμπιστοσύνη και την ανάπτυξη. Η άλλη διάσταση που πρέπει να δούμε είναι ότι η αλυσίδα της αξίας σήμερα ε, είναι πολύ πιο περίπλοκη σε σχέση με το παρελθόν. Οπότε αυτά τα μέτρα έχουν τελείως διαφορετικό αντίκτυπο ανάλογα με την παγκόσμια λυσίδα παραγωγής και αξίας. είναι αυτές οι επιδράσεις πολύ σημαντικές και πιθανώς σοβαρές. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το τελικό άθροισμα όλων αυτών, αλλά θα ξέρουμε ότι θα είναι μεγάλο και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προετοιμαστούμε. Αν όσα έχουν ανακοινωθεί ισχύσουν και όσα ακολουθήσουν μετά θα είναι πολύ σοβαρά. Τέλος, αναφέρατε τον κίνδυνο μιας υψηλής ανατίμησης, ε, μιας υψηλής ε, με συγχωρείτε, ε, των τιμών των στοιχείων του ενεργητικού. Είναι κάτι το οποίο παρακολουθούμε. Οι τράπεζες συνολικά φαίνεται ότι είναι προετοιμασμένες για μια γρήγορη αύξηση των επιτοκίων υπό την έννοια ότι οι προσωμιώσεις που έχουμε κάνει, τα μοντέλα που έχουν κάνει και οι τράπεζες δείχνουν ότι όταν ανεβαίνουν τα επιτόκια ανεβαίνει και το καθαρό περιθώριο των επιτοκίων αν και, οπότε συνολικά οι τράπεζες είναι σε καλύτερη θέση αν και βέβαια εξαρτάται και το ποιο είναι το χαρτοφυλάκιό τους αλλά θα ε, πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί και να μην εφησυχάζουμε, γιατί τα μοντέλα στα οποία βασίζονται αυτά τα συμπεράσματα είναι μοντέλα που σχεδιάστηκαν μετά από μία περίοδο πολύ χαμηλών επιτοκιών και υποθέτουν ότι η προσαρμογή των ε, επιτοκίων χορηγήσεων θα είναι πιο αργή από την ε, προσαρμογή των επιτοκίων δανεισμού, κάτι το οποίο δεν είναι απαραίτητα αλήθεια. Ο Νότς Μαριάς. going to speak in Greek. Ευχαριστώ. Ε, κύριε Πρόεδρε, πριν από λίγες μέρες ήρθε στη δημοσιότητα μία μελέτη των οικονομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με θέμα μαθαίνοντας για τους δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές fiscal multipliers κατά τη διάρκεια της κρίσης του ευρωπαϊκού χρέους. Την έχω εδώ αυτή τη μελέτη, η οποία λίγος πολύ λέει, κύριε Πρόεδρε, ότι η απόφαση και του Eurogroup και της Τρόικας να υπάρξει μια σκληρή δημοσιονομική πολιτική και κυρίως να μειωθούν οι δαπάνες σε χώρες που μπήκαν σε μνημόνια όπως η Ελλάδα, είχε δυσμενή αποτελέσματα, διότι έγινε λάθος εκτίμηση στον δημοσιονομικό πολλαπλασιαστή. Επομένως οι συνέπειες ήταν αρνητικές, οι χώρες βυθίστηκαν σε ακόμη μεγαλύτερη κρίση και φυσικά στην Ελλάδα είχαμε στρατιές ανέργων, είχαμε χιλιάδες φτωχούς, μείωση μισθών, συντάξεων κλπ. Το ερώτημα είναι ότι εφόσον ακόμη και οι οικονομολόγοι που δούλεψαν για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το δέχονται το λάθος το οποίο έγινε. Δηλαδή το λάθος των πολλαπλασιαστή. Ένα λάθος που είχε αναγνωρίσει και το Δούνου του από το 2015. Και επειδή η ΕΚΟΥΤΟΥ συμμετείχε έντονα στη διαμόρφωση αυτών των προγραμμάτων και στην παρακολούθηση. Και επειδή κύριε Πρόεδρε εδώ, σε αυτή την αίθουσα και εγώ ίδιος, πολλές φορές σας είχα θέσει το ίδιο ερώτημα. Ότι κάνετε λάθος στην εκτίμηση ότι κακώς προχωρείται σε μια πολιτική ω Τρόικα που επιβάλλει μείωση των δαπανών, διότι έτσι οδηγεί σε μεγαλύτερη ύφεση στη χώρα. Τώρα λοιπόν που έρχονται αυτά τα πράγματα στη δημοσιότητα και έχουμε δει και τις δυσμενείς συνέπειες, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι διατεθειμένη να αποζημιώσει την Ελλάδα για την τεράστια ζημιά την οποία έχει υποστεί η δική της οικονομία. Διότι έχουμε, όπως γνωρίζετε κύριε Πρόεδρε, φτωχοποίηση του ελληνικού λαού και διάλυση φυσικά της ελληνικής οικονομίας. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε να πω κάτι. Το έγγραφο που αναφέρατε δεν είναι η επίσημη θέση της ΕΚΤ είναι το πρόγραμμα που απορρέπει την έρευνα. Δημοσιεύεται υπό την ευθύνη των συγγραφέων του εγγράφου. Το αναφέρει εκεί, το αναφέρει κάτω, σαν υποσημείωση. Εν γέννη, να σας πω το εξή. Η ΕΚΤ θα προβεί σε μια αξιολόγηση της όλης εμπειρίας εφαρμογής των προγραμμάτων μας και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Αυτό είναι σίγουρο. Έχετε όμως υπόψη ότι η καλύτερη συνεισφορά που έκανε η ΕΚΤ στην Ευρωζώνη ήταν να πετύχει τη σταθερότητα των τιμών. Και θα σταματήσω εδώ και θα επανέλθουμε από αυτού όταν θα έχουμε τη δική μας αξιολόγηση των προγραμμάτων. Δεν θα βασίσω τα συμπεράσματά μου σε ένα πρόγραμμα που είναι αποτέλεσμα έρευνας, παρόλο που κάποια από τα συμπεράσματα που αναφέρεται στον αφορά τον πολλαπλασιαστή, για τους πολλαπλασιαστές που ήταν διαφορετικοί σε παρατεταμένες υφέσεις και ε, σε περίπτωση φορολόγησης σε διάφορες περιόδους, δεν είναι κάτι μοναδικό σε αυτό το έγγραφο. Mr. Chairman, I will... Δεχθώ δηλαδή ότι αφού εξετάσετε κι εσείς ως Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα δεδομένα, λάβετε υπόψη και αυτή τη μελέτη των οικονομολόγων, εάν αποδειχθεί ότι πράγματι έχουν γίνει λάθη από την πλευρά της Τρόικας, να το εκλάβω πλέον ότι θα εξετάσετε ως Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την αποζημίωση της Ελλάδος για τη ζημιά που έχει υποστεί. Thank ε, you. As I have some more seconds. Αντιλαμβάνομαι, αντιλαμβάνομαι ότι έρχεστε σε πολύ δύσκολη θέση, αλλά βεβαίως εάν και εφόσον... Okay. So, the next question is as follows. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι είναι δύσκολη θέση της ΕΚΤ να απαντήσει, αλλά δεν πειράζει. Θα το δούμε στο μέλλον. Το ερώτημά μου έχει να κάνει τώρα με τις συντάξεις στην Ελλάδα. Επειδή συμμετέχετε στην Τρόικα, και ήρθατε το Σεπτέμβριο στην Ελλάδα. Και έχει αποδειχθεί ότι δεν χρειάζεται να μειωθούν οι συντάξεις. If you don't interrupt me, and if you give me the time for the socialist group six minutes you gave before, I will finish. Okay. Οπότε, κύριε Πρόεδρε, finally, my question, my question for you in, in Greek. I mean, I know, I know the answer. Ε, το ερώτημα είναι εσείς επιμένετε στη μείωση των συντάξεων παρότι δεν χρειάζεται να μειωθούν οι συντάξεις διότι έχει αποδειχθεί ότι δεν απαιτείται μείωση των συντάξεων με βάση τους δημοσιονομικούς όρους σήμερα στην Ελλάδα. Ευχαριστώ. Uh, the, the ECB όταν εξέτασε την συμμετοχή της στο πρόγραμμα προσφάτως κατέληξε στο ότι χρειαζόμασταν ένα διαφορετικό πλαίσιο λειτουργίας, δηλαδή να ασχοληθούμε με την μακροοικονομική και χρηματοπιστωτική πτυχή της οικονομίας, οπότε δεν θα πούμε πια τίποτα άλλο ε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για συντάξεις, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ιδιωτικοποιήσεις και πολλά πράγματα για τα οποία ομολογουμένως και τα τελευταία χρόνια είπαμε κάτι δευτερευόντως. Ναι, ναι. Να σας πω κάτι λίγο ως πρόεδρος της αρμόδιας ομάδας εργασίας. Όπως ξέρετε, το 1% των μέτρων για τη συντάξη συν άλλο 1% ως φορολογικά μέτρα τα ζήτησε το ΔΝΤΑΦ και κανένα θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χαίρεται ιδιαίτερως γι' αυτό, οπότε η ερώτηση αυτή πρέπει να απευθυνθεί σε άλλους. Και το, το, δεν ήταν προς συζήτηση. Ο κύριος Μαριάς, ναι, αυτό θα το δει το, το Eurogroup και πρέπει το Κοινοβούλιο να επιμείνει σε μη περικοπή. Λοιπόν, δεν έχετε άλλο τον λόγο. Κύριε Βόλφ, περνάμε στο KTI. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Ντράγκη. Χαίρομαι που ήρθατε σε αυτή την Επιτροπή. Το σύστημα μετά το Bretton Woods ε, θα έλεγα ότι ε, παλεύει. Βλέπουμε και την κρίση του 1970, τις πετρελαϊκές κρίσεις, ε, την κρίση του 80. Οι κρίσεις λοιπόν έρχονται όλο και συχνότερα. Βεβαίω το ευρώ δημιουργήθηκε ακριβώς λόγω αυτού του σενάριου γιατί είχε αποσυρθεί από τον χρυσό κανόνα το δολάριο. Λοιπόν, κοιτάω εδώ πέρα κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Το ότι έχουμε ένα παράλληλο σύστημα με τους ισολογισμούς των κεντρικών τραπεζών, η απόδοση των ομολόγων ως ποσοστό του ΑΕΠ που είναι σε ιστορικά αρνητικά επίπεδα, έχουμε ακραία επίπεδα παγκόσμιων ανισορροπιών και βεβαίως αυτό επηρεάζει και την χαμηλή οικονομική ανάπτυξη. Δύο ερωτήσει, λοιπόν. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει κάνει κάποιον χοντρικό υπολογισμό το πόσο επηρεάζουν οι μετοχέ και τα ομόλογα και η τυχόν υποτιμησή τους και δεδομένου του ότι μάλλον έρχεται και άλλη μια κρίση πια μέσα έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεδομένου του ότι τα περισσότερα τα έχει εξαντλήσει την δεκαετία που μας πέρασε. Σας ευχαριστώ. Έχουμε κάνει προσωμιώσεις ε, για τα πιθανά αποτελέσματα μιας ε, έντονης ε, αλλαγής της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού. Και το είπα και πριν, είναι πολύ ισχυρότερε σήμερα οι τράπεζες. Υπό μια έννοια μπορούν να αντέξουν κάποια από αυτά τα αποτελέσματα, αλλά είπα να μην είμαστε και υπερβολικά αισιόδοξοι από λόγο μοντέλων που βασίστηκαν σε μία μακρά περίοδο χαμηλών επιτοκίων, γιατί οι παράμετροι αυτών των μοντέλων επηρεάζονται από την εξαιρετική κατάσταση των τελευταίων δεκαετών. Αλλά και πάλι η περιορισμένη αυτή εμπιστοσύνη δεν εκτείνεται οπωσδήποτε στον τομέα, τον σκιώδη, τον σκιώδη τραπεζικό τομέα, όπου δεν έχουμε τόσο μεγάλη διαφάνεια και όπου τα ιδρύματα είναι μεγάλα, περίπλοκα και διασυνδεδεμένα και έχουν αποκτήσει μεγάλη σημασία και κάνουν ε, επιτελούν ε, τις λειτουργίες των τραπεζών πολύ περισσότερο σήμερα από ό,τι στο παρελθόν. Η ΕΚΤ, λοιπόν, οπότε σε γενικές γραμμές ε, κοιτάμε, παρακολουθούμε. Συγχωρείτε. Λοιπόν, η ΕΚΤ η ίδια έχει τα μέσα για να ακολουθήσει ακριβώ μια πολιτική σταθερότητα στον τιμών. Δεν μα λείπουν τα μέσα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους ε, και τον κύριο Ντράγκη για την έντονη και ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση, τον νομισματικό διάλογο. Μπορούμε τώρα να περάσουμε λοιπόν στο επόμενο θέμα τη συζήτησή μα και θα δώσω τον λόγο στον Brian Hayes. Σα ευχαριστώ κύριε Τρέπη. <coughs> Ευχαριστώ συνάδελφοι. Πάμε στο επόμενο σημείο της ημέρας διάταξης. Πρόθεση της χρήσης της αγοράς των αγορών για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο συνάδελφος Σάντερ έχει το λόγο να μας μιλήσει για το θέμα. Η Σάντερ, μάλλον. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας, είναι πάνω από 99% των επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικές για την ανάπτυξη στην επικράτειά μας, διότι δημιουργούν θέσεις απασχόλησης και δημιουργούν κυρίως βιώσιμες θέσεις εργασίας και ποιοτικές θέσεις. Είναι παρούσες όλους τους τομείς και σε μελλοντικού τομείς όπως η βιοτεχνολογία, ψηφιακός τομέας, η υγεία, η μηχανολογία εχμής, οι επικοινωνίες. Αυτές οι μικρές επιχειρήσεις που σήμερα πραγματικά είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εκείνες ίσως θα είναι γίγαντες αύριο. Συνεπώς, σαν συνομοθέτες, θα πρέπει να λάβουμε καλύτερα υπόψη τις ιδιαιτερότητες των εν επιχειρήσεων και να εφαρμόσουμε την αρχή της αναλογικότητας στο συχνότερο δυνατόν. Μετά την οικονομική κρίση του 2008, Είχαμε καταιγισμό εγγράφων που ρύθμισαν το χρηματοστατικό τομέα και που εις βάθος βελτίωσαν την αντοχή του συστήματος και τη λειτουργία του. Έχουμε ένα χρηματοστατικό τομέα πιο ασφαλή, αλλά λόγω κανόνων που είναι αυστηροί, πολύ αυστηροί καμιά φορά, δεν επιτρέπει τη χρηματοδότηση οικονομίας όπως θα έπρεπε. Σήμερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νεοφυείς επιχειρήσεις αλλά επίσης και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις έχουν δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοδότησή τους. Η ποικιλομορφία των επιχειρήσεων απαιτεί πολύ διαφορετική χρηματοδότηση και στα πλαίσια της Ένωσης των Κεφαλαγορών πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποιες πρωτοβουλίες με στόχο ποικιλομορφία όσον αφορά την πηγή χρηματοδοτήσεως των επιχειρήσεων αλλά πρότεινε και χρηματοδότηση πιο καλά προσαρμοσμένη Αυτές οι νομοθετικές προτάσεις οι με την αγορά που βοηθά την ανάπτυξη των επιχειρήσεων είναι κάτι που εξεργαστήκαμε και είναι μια καλή δυνατότητα να προσαρμόσουμε τους χρηματοπιστωτικούς κανόνες που ανέφερα ε, στην επικαιρότητα. Όταν το πακέτο MIFID 2 MIFIR υιοθετήθηκε το 2014, οι διατάξεις επέτρεπαν τη δημιουργία πλατφορμών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, που αποτελούν την αγορά για την ανάπτυξη αυτών. Το κείμενο πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μειώσει το διοικητικό και ρυθμιστικό πλαίσιο ε, για να χαλαρώσει το πλαίσιο για τις ε, επιχειρήσεις αυτές που έχουν εισαχθεί στην αγορά κεφαλαίων. Λοιπόν, έχουμε και το προσπέκτους ε, που αναθεώθηκε πρό, ε, πρόσφατα και τον νέο κανονισμό. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά την άποψή μου, ε, που έγινε, είναι μια ευκαιρία, πρέπει να την αρπάξουμε και οι χαλαρώσει του πλαισίου που προτείνονται ακολουθούν την καλή κατεύθυνση. Πιστεύω όμως ότι μπορούμε να προχωρήσουμε πιο πέρα και εν αυτή τη ενία πρότεινα κάποιες τροπολογίες. Στο σχέδιο της εκθέσεως που συζητούμε σήμερα, ε, θα ήθελα να προτείνω κάποιες ε, βελτιώσεις που έχουν στο στόχο να επιτρέπουν σε περισσότερες επιχειρήσεις να μπορούν να μπουν σε αυτή την αγορά ανάπτυξης τροποποιώντας το όριο που καθορίζει μια μικρομεσαία επιχειρήση στο MIFID αλλά και στο προσπέκτους. Αυτές οι αλλαγές θα πρέπει να ε, έχουν στόχο τις εισηγμένες αυτές ε, μικρόμεσες επιχειρήσεις. Θα πρέπει και οι διοικητικοί περιορισμοί όσον αφορά τους κανόνες για κατάχρηση αγοράς να χαλαρώσουν, όσον αφορά τη δημοσίευση καταλόγων ατόμων που συνδέονται ε, με τη διαχείριση επιχειρήσης ή τους κανόνες για τη δημοσιοποίηση απορρίτων πληροφοριών, εμπιστευτικών πληροφοριών. Το σχέδιο εκθέσεως έχει στόχο τους επενδυτές προτείνεται να εξαιρεθούν ιδιωτικέ τοποθετήσει από τη δημοσκόπηση τη αγορά και από την αγορά τη ανάπτυξη και από την ρυθμιζόμενη αγορά. Λοιπόν, οι ιδιωτικέ αυτέ επενδύσει λόγω των ε, γενών χαρακτηριστικών δεν απαιτούν κάποιο περιορισμό. Θα πρέπει να έχουμε ένα όραμα πιο σφαιρικό και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει εντολή να εξολογήσει κατά πόσο οι χαλαρώσεις ή τροποποίησεις αυτές θα μπορούν να εφαρμοστούν στο προληπτικό πλαίσιο των επενδυτών και στο MIFID 2 και MIFIR, ούτω ώστε να γίνουν ιδέωσες προσαρμογές για τις νομικές επιχειρήσεις. Με άλλα λόγια, σκοπός είναι να ανοίξουμε νέες πηγές χρηματοδοτήσεως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να απλουστεύσουμε τους κανόνες Αυτά λοιπόν προτείνονται στην έκθεσή μου κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα να πω πάνω απ' όλα ότι χαίρομαι που ακούω τις διάφορες προτάσεις, συστάσεις, ε, να ακούσω μάλλον, θέλω να ακούσω με χαρά τις συστάσεις και προτάσεις των συναδέλφων. Αυτά και ευχαριστώ.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 να σας πω βέβαια πως ε, επειδή εκλέγεται στα Wesley Midlands όπου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της τοπικής οικονομίας είναι ιδιαίτερα, ε, αισθάνεται ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το φάκελο αυτό και κυρίως για το πώς θα μπορούσαμε να χρηματοδοτήσουμε τις μικρομεσαίες. Αυτό αποτελεί και μία από τις βασικές τους ανησυχίες. Πιστεύει λοιπόν πως η πρωτοβουλία αυτή, η οποία έχει ως στόχο τη διεύρυνση ε, στις πηγές χρηματοδότησης, είναι καλοδεχούμενη, αρκεί, αρκεί κάποιες ασφαλιστικές δικλίδες να τοποθετηθούν στο κείμενο. Δηλαδή να βρούμε μια ισορροπία αφενός μεταξύ της μείωσης της γραφειοκρατίας έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη ανάπτυξη και πρόσβαση στη χρηματοδότηση και αφετέρου να έχουμε επαρκή προστασία των επενδυτών. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να δημιουργηθούν με τον κατάλληλο τρόπο και για όλα αυτά και για το ισοσύγιο, και για την κεφαλαιοποίηση και για τα κατόφλια και για τα όσα προτείνει η συγγήτρια. Θα τα ξαναδεί με προσοχή και θα τα σχολιάσει. Καλό είναι να γίνει και μια αξιολόγηση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις μιας πρότασης σαν αυτή που καταθέτει η συγγήτρια. Δηλαδή, το κατόφλι ε, για τον ορισμό για το μικρομεσαία επιχείρηση και πώς αυτό αλλάζει από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Γιατί για το μέγεθος πάντα προκύπτει η ίδια συζήτηση. Δηλαδή, οι μικρομεσαίες μπορεί να μην ορίζονται επαρκώς ε, ήταν μπορούν όλες να περιγραφούν με τον ίδιο τρόπο. Παρ' όλα αυτά χρειάζεται κάποιος ορισμός στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για να βρούμε τη σωστή η νομοθεσία και για τον κανονισμό για το προσπέκτος και, για την, τον κανονισμό για την ε, ε, καταπάτηση του κανονιστικού πλαισίου η Νίνα Γκίλ λέει πως είναι θετικά όλα αυτά αρκεί να μην επηρεαστεί η προστασία των ε, επενδυτών. Και σε αυτά τα πλαίσια θα χαρεί και εδώ να γίνει μια αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις προτάσεις της εισηγήτριας. Δηλαδή, για το να αλλάξουμε από τα τρία στα δύο έτη την περίοδο κατά την οποία έχουν πρόσβαση οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αυτές τις αγορές. Εκτός από αυτές τις παρατηρήσεις, όπως πάντα, και όπως οποιοδήποτε κανονικός ευρωβουλευτής είναι ε, πάντα πρόθυμη να συζητήσει με την εισηγήτρια τα θέματα που του αφορούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ Περβάος. Εκ μέρους της ECR. Δεν βλέπω κάποιον. Δεν βλέπω την Εύα. Αν έρθει αργότερα θα της δώσω το λόγο. Από τους φιλελεύθερους. Κανείς. πράσινη. Ο Φιλίπ Λαμπέρ. Να βρούμε κάποιον από την ΚΟΕ. Εκτός μικροφώνη, κυρία Μπερές. Λοιπόν, όλοι καταλήγουμε στα συμπεράσματά μας. Η FTD. Όχι. Να περάσουμε λοιπόν στη διαδικασία κάτι διά Θέλει κάποιος συνάδελφος κάτι να πει. Νομίζω ότι μας έδωσαν τη λάθος χρονοθυρίδα για το θέμα αυτό. Θα ήθελα λοιπόν εσύ ως εισηγήτρια να απαντήσεις αν δεν υπάρχει άλλος συνάδελφος ο οποίος να έχει σχόλια. Ε, αν. Καταλήγω στο εξή συμπέρασμα, κύριε Πρόεδρε, πως το κείμενο αυτό θα πρέπει να είναι πραγματικά Α, με συγχωρείτε. Δείχνω πως είμαι άπειρος, δεν έχω δώσει το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κομισιόν, θέλετε να απαντήσετε σε αυτά που ακούστηκαν. Uh, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την εισηγήτρια που εργάστηκε για αυτό τον τόσο σημαντικό φάκελο και για εμάς και για την συμπλήρωση ε, του όλου έργου μέχρι το Δεκέμβριο. Οπότε σας ευχαριστώ κυρία εισηγήτρια. Δεύτερον, Και επίση θα θέλαμε να την ευχαριστήσουμε για κάποιες από τις προτάσεις, θα τι κοιτάξουμε και κάποιες από τι τροπολογίε ίσως τελικά ε, βελτιώνουν την πρόταση της δική μα, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακόμα βρισκόμαστε βέβαια σε πολύ πρώιμο επίπεδο των αναλύσεων του θέματος που έχουμε κάνει. Λυπόμαστε πολύ. Φτάσαμε λίγο καθυστερημένα, οπότε ε, μπορείτε να μου υπενθυμίσετε τι ερωτήματα έκανε η εισηγήτρια, γιατί δεν είχαμε μπει στην αίθουσα την ώρα που μίλαγε. Και βεβαίω αν κάτι στρέφεται προς εμάς, θα απαντήσουμε μεγάλη χαρά. Okay, so... No one else is going to take the floor at stage. άλλος αγορεύει, που λέτε. Λοιπόν, προθεσμία για υποβολή τροπολογιών, 9 Οκτωβρίου, 9 Οκτωβρίου, συζήτηση από αυτόν 19 Νοεμβρίου, ψηφοφορία στην ΕΚΟΝ 3η Νοεμβρίου. Α, Δεκεμβρίου, γι' αυτό Δεκεμβρίου. Αν... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμπεραίνω ότι το κείμενο οδηγεί σε συνένεση. Δεν είδα να υπάρχουν παρατηρήσεις από τις άλλες πολιτικές ομάδες, εκτός από το σχόλιο των σοσιαλιστών. Οπότε κατανόησα αυτό που είπε η κυρία Μπερές με κάποιες ερωτήσεις που απευθυνθούν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα περιμένουμε κάποιες απαντήσεις. Αυτό ζητούν οι σοσιαλιστές. Κυρίως επί κάποιων προτάσεων και κυρίως επ' αυτής που αφορά το κατόφλι που επιτρέπει σε περισσότερες μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις να ωφεληθούν, να έχουν πρόσβαση σε αυτή την αγορά της ανάπτυξης. Αδιαφυσβήτητα θα έχουμε τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις εμβαθύνοντας στο θέμα αυτό με τους κοιόδης ηγητές. Ελπίζω. Και θα χαρώ να συνεργαστούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Αν. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι θα λάβετε πολλές τροπολογίες και θα έχουν και την ευκαιρία να μιλήσουν, αλλά είναι απογοητευτικό να μην είναι εδώ ο κόσμος για την συζήτηση. Για βεβαίω πρέπει να πούμε ότι μπορεί και να μην έχουν καμία αντίρρηση για το κείμενο σου. Η προθεσμία για τροπολογίες ε, είναι όπως είπα και σκοπεύουμε να ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας ε, γύρω στις 3 Δεκεμβρίου. Λοιπόν, διάλειμμα ολίγων λεπτών καθώς περιμένουμε το σημείο 6. Μείωση του αντικτύπου ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον. Διάλειμμα 15 λεπτών. Ευχαριστώ. So, colleagues, welcome back to our next item. It's point number in our... Λοιπόν, συνάδελφοι, περνάμε στο επόμενο θέμα της και διάταξης. Μείωση του αντικτύπου ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον. Θα το ψηφίσουμε αυτό σήμερα, αμέσως μετά το σημείο 7. Και έχουμε 120 τροπολογίες. 36 εκ των οποίων είναι από την εισηγήτρια η οποία έχει αμέσως τον λόγο η κυρία Κάπελ η συνάδελφος από την Αυστρία που θα μας πει τώρα πώς έχουν τα πράγματα Μπάρμπαρα Λοιπόν, τέλος πάντων ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή και να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές Έγινε πολλή δουλειά σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. 3 Σεπτεμβρίου μας ενημέρωσε η γραμματεία και σήμερα είναι 24. Ψηφίζουμε ήδη, οπότε είχαμε πάρα πολύ δουλειά να κάνουμε και να ευχαριστήσω πραγματικά τις ομάδες και τους κοιόδης ηγητές. Ξέρουμε ότι χωρίς τους συνεργάτες μας δεν θα τα καταφέρναμε. Να πω επίσης ότι ήμουν και σκιώδη συγγήτρια στην Ήτρε για την γνωμοδότηση για τα πλαστικά, η οποία ψηφίστηκε σήμερα και πήγανε πολύ θετικά τα πράγματα, είχαμε μεγάλη πλειοψηφία και να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές ειδήσει στα ΜΜΕ στην Αυστρία σχετικά για τα πλαστικά και η Κομισιόν έχει κάνει την πρόταση να απαγορευτούν ε, σταδιακά τα πλαστικά μιας ε, χρήσης και είπαμε στις συναντήσεις των σχεδόν εισηγητών ότι πρέπει να δούμε και την αρχή της αναλογικότητας γνωρίζοντας ότι ένα μεγάλο κομμάτι των 50.000 ε, των επιχειρήσεων που ασχολούνται σε αυτόν τον τομέα είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να περάσουν βεβαίως σε μια νέα ρύθμιση ε, να μπορέσουν βεβαίως να κάνουν και την απαραίτητη σημανσή των διασπόμενων υλικών αλλά να έχουν πρώτα απ' όλα την ευκαιρία και πρώτον τον χρόνο να προετοιμαστούν και δεύτερον την ικανότητα να έχουν και περισσότερα κονδύλια για έρευνα και ανάπτυξη στον πολύ καινοτόμο αυτόν τομέα για να αυξήσουν έτσι την ανταγωνιστικότητά τους. Ταυτόχρονα βεβαίως πρέπει να ενημερώσουμε και τους ανθρώπους ε, για την ανακύκλωση, την επαναχρησιμοποίηση, την κύκλική οικονομία και πρέπει να το δούμε και παγκοσμίως γιατί γνωρίζουμε ότι 80% της ρήπανσης από πλαστικά στις θάλασσες δεν προέρχεται από την Ευρώπη αλλά από άλλες χώρες αναπτυσσόμενες και τις ΗΠΑ. Οπότε πρέπει να δραστηριοποιηθούμε σε παγκόσμιο επίπεδο και βεβαίως πάντα ακολουθώντας την αναλογικότητα να έχουν την δυνατότητα επιχειρήσει να είναι ενήμερες. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε την εισηγήτριά μας. Περνάμε τώρα στους σκιωτισηγητές. Ρωμάνα Τόμσον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ την κυρία Κάπελ για την συνεισφορά της Πράγματι ήταν πολύ αποτελεσματική η συνεργασία μας, είχαμε ελάχιστο χρόνο, όμως καταφέραμε να συμφωνήσουμε στα περισσότερα σημαντικά ζητήματα που εκκρεμούσαν. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους συναδέλφους της ALDE και του ECR, διότι ήταν πολύ πρόθυμοι να συνεργαστούν. Η οδηγία που αφορά τη μείωση το αντιχτύπου κάποιων προϊόντων πλαστικού ε, είναι κάτι πολύ θετικό για το περιβάλλον μας και για το μέλλον μας. Εγώ θα εξέφρασα την ευχή και το Ευρωκοινοβούλιο να αναγνωρίσει τη σημασία που έχει αυτή η ευκαιρία που παρουσιάζεται για τη βιομηχανία μας. Αυτό είναι κάτι που πολλές φορές το λησμονούμε. Οι μικρές και οι μεσαίο μεγέθους επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας είναι οι επιχειρήσεις που μπορούν να προσαρμοστούν πολύ γρήγορα στις νέες συνθήκες της αγοράς. Ελπίζω ότι αυτή η οδηγία δεν θα περιορίσει τις εργασίες τους, αλλά θα τους δώσει ένα προσανατολισμό, ε, θα τις κατευθύνει προς τη σωστή κατεύθυνση για να αναπτυχθούν. Θα είναι κάτι επωφελές και για αυτές και για μας. Όπως ανέφερε και η Μπάρμπαρα, η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση είναι πάρα πολύ σημαντικό και εδώ έχουμε μείνει κάπως πίσω δεν χρησιμοποιούμε αρκετά μέτρα για την ευαισθητοποίηση του κόσμου, κυρίως να γίνει κατανοητό ότι δεν είναι ένα πρόβλημα που αφορά μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται σε παγκόσμιο επίπεδο κάποια προσέγγιση. Τα προβλήματα με τα απόβλητα από πλαστικό δεν περιορίζονται στα σύνορα μιας χώρας. Θα πρέπει να περιορίσουμε τα πλαστικά μιας χρήσεως σε όλους τους τομείς της ζωής, όπου τέτοια προϊόντα δεν είναι βασική σημασίας. Έτσι μπορούμε να υποχρεώσουμε τους παραγωγούς ε, σιγά σιγά να σταματήσουν να παράγουν αυτά τα προϊόντα. Βέβαια θα πρέπει ταυτόχρονα να τους ε, ευαισθητοποιήσουμε και να τους βοηθήσουμε να αναπτύξουν καλύτερα νέα προϊόντα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ρωμάνα. Δεν έχουμε κανέναν από τους σοσιαλιστές, ε, τουλάχιστον σκιώδη. ECR. Λούκε. Ευχαριστώ, Μπράιν. Ευχαριστώ την κυρία Κάπελ, την ε, εισηγήτρια για την γνωμοδότηση αυτή. Θα επιβεβαιώσω αυτό το οποίο είπαν οι συνάδελφοι. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή και αποτελεσματική συνεργασία. Να ευχαριστήσω λοιπόν τους εκπροσώπους ε, του ΕΛΚ της Άλντε και βεβαίως την κυρία Κάπελ. Είναι πολύ σημαντικό το ότι ε, ανέλαβαν οι κέντρο δεξιές ε, δυνάμεις εδώ στο Κοινοβούλιο το θέμα αυτό, το οποίο δεν ήθελαν οι σοσιαλδημοκράτες. Ε, φαίνεται λοιπόν, ίσως ποιος ενδιαφέρεται ουσιαστικά. Λοιπόν, Θεωρώ ότι τελικά βρήκαμε μια καλή λύση για το θέμα αυτό χωρίς να οδηγηθούμε σε υπερβολική επιβάρυνση των επιχειρήσεων. Και ακριβώς ε, ε, φροντίσαμε να μην υπάρχει κάποια στρέβλωση του ανταγωνισμού εις βάρος των εγχωρίων ε, επιχειρήσεων που παράγουν εντός της Ένωσης σε σχέση με όσων παράγουν εκτός ε, και εξάγουν στην Ένωση. Πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το θέμα γιατί κάποιες προτάσεις της Κομισιόν δεν το έχουν λάβει επαρκώς υπόψη. Και θεωρώ λοιπόν ότι μπορούμε να έχουμε πολύ ψηλέ προσδοκίες από την νομοθεσία αυτή την οποία θα ψηφίσουμε απόψε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχουμε τον Βέλγο συνάδελφο, την κυρία Βερνίκ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα... Ε, θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για όσα κάνατε και όσοι πήρατε μέρος ήσασταν πάρα πολύ επικοδομητικοί. Γι' αυτό λοιπόν με πεποίθηση μπορώ να σας πω πως στηρίζουμε πλήρως αυτή την πρόσταση. Τα πλαστικά στο περιβάλλον μας είναι ένα πρόβλημα που διωγγώνονται με αρνητικές συνέπειες για τους ανθρώπους, τα ζώα και το περιβάλλον. Αυτά είναι σαφές. Η λύση όμως για το πρόβλημα δεν είναι μόνο στα χέρια των παραγωγών. Έχει και ο καταναλωτής ο οποίος θα χρειάζεται να αλλάξει νοοτροπία. Και προς αυτή την κατεύθυνση είμαι πραγματικά ντυμένη για να συζητήσουμε αυτή την έκθεση γιατί είναι 100% ε, ανακυκλωμένο από πλαστικά μπουκάλια το φορεμά μου και το 30% από αυτά τα μπουκάλια που χρησιμοποιήθηκαν συλλέχθηκαν από τον ωκεανό. Ας ανακυκλώνουμε λοιπόν και ας ανακυκλώνουμε όλο και περισσότερα έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε το μέλλον. Και συγχαρητήρια για το ότι είστε μοντέλο σήμερα για τους υπόλοιπους από εμά σε επίπεδο ενδυματολογικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από την ΚΟΕ ποιος θέλει να πάρει το λόγο. Ωραία, περνάμε στο Catch the Eye. Ο κύριος Φέρμπερ, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που σας βλέπω στην έδρα. Έχω κάποιες ερωτήσεις, γιατί έχω καταθέσει κάποιες τροπολογίες. Υπάρχουν κάποιες ουσίες που μοιάζουν με το πλαστικό, αλλά είναι διασπόμενες ε, φυτικές ουσίες που είναι αρκετά σκληρές, αλλά μετά από τρεις ή έξι μήνες ε, διαλύονται και μπορούν να πεταχτούν στο λόφο της ε, κομποστοποίησης. Γι' αυτό μου προξενεί ε, εντύπωση το ότι δεν αναφέρθηκαν αυτά από την εισηγήτρια. Θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι η αιτία. γιατί μιλάμε για μη διασπόμενα πλαστικά, πολυπροπυλένιο κτλ. να απαγορευτούν. Εντάξει. Αλλά άλλα προϊόντα τα οποία δεν είναι πλαστικά αλλά ομοιάζουν θα καλύπτονται αυτόν τον προϋπολογισμό. Ενώ έχουμε εναλλακτικέ ε, που παραγόνται στην Ευρώπη με βάση φυτικές πρώτες Οπότε θα ήθελα να ληφθούν υπόψη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραιότατα. Υπάρχουν άλλα αιτήματα για το Catch the Eye πριν ξαναδώσω τον λόγο στην εισηγήτρια. Όχι, Μπάρμπαρα, λοιπόν, εάν μπορείτε να απαντήσετε δεδομένου το ότι είχαμε και πολύ σημαντική πρόοδο από τους συμμετέχοντες. Κοιτάξτε, ε, κάποιο οπωσδήποτε καλύπτονται δηλαδή θα εξαιρεθούν από την απαγόρευση τα διασπόμενα προϊόντα και πρέπει να υπάρξει μια ρύθμιση η οποία δεν υπάρχει βεβαίως ακόμα αλλά εγώ δεν βλέπω κάποιον λόγο για την απαγόρευση των διασπόμενων υλικών. Ούτως ή άλλως νομίζω δεν θα υπάρξει τέτοια απαγόρευση στο πλαίσιο της αναλογικός, αλλά το είπαν και οι είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα γιατί όπως είπαμε κάθε χρόνο έχουμε 500.000 τόνους ε, πλαστικά απορρίμματα που καταλήγουν στους ωκεανούς και πρέπει να δούμε αυτές τις απειλές ε, για την ανθρώπινη υγεία. Και προξενή εντύπωση που δεν ενδιαφέρεται ο κόσμος. Α, τέλος πάντων έτσι είναι η δημοκρατία. Ελπίζω να έρθουν τουλάχιστον για την ε, ψηφοφορία. Προσπαθήσαμε λοιπόν να συνεννοηθούμε και με την Επιτροπή ΕΝΒΙ και με όσους ασχολούνται με αυτό το θέμα και καταφέραμε ομαδικά να προετοιμάσουμε θα έλεγα μια καλή γνωμοδότηση και όπως είπε και ο κύριος Φέρμπερ δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αν υπήρξε μια πρώτη αρνητική αξιολόγηση της ε, τροπολογίας του, λυπούμε. Μπορεί βεβαίως να την ε, δούμε θετικά. Τα μη διασπόμενα πρέπει να αντικατασταθούν. Υπάρχουν ήδη καινοτόμα προϊόντα. Και βεβαίως δεν θέλουμε να εμποδίσουμε τα διασπόμενα. Σας ευχαριστούμε. Μπάρμπαρα, περνάμε στο σημείο 7. Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου. Περνάμε κατευθείαν στον συνάδελφο τον Μιγγέλ Βιέγκας από την ΚΟΕ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πω στα γρήγορα γιατί ξέρετε πως χρειαστήκε να τρέξουμε γιατί οι προθεσμίες δεν ήταν θετικές μέσα στο καλοκαίρι χωρίς να προλάβουμε να συζητήσουμε όπως θα είχαμε προτιμήσει. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια γιατί η δική μας αντιμετώπιση του θέματος είναι πως γενικά εδώ αντιμετωπίζουμε την οδηγία αυτή συνενετικά και προσπαθούμε να βρούμε τον κοινό παρανομαστή ο οποίος θα μας επιτρέψει να καταλήξουμε σε μια τελική πρόταση ε, η οποία θα εκπροσωπεί όλους τους συναδέλφους. Αυτή είναι η προσέγγιση την οποία ακολουθήσαμε. Δεν το καταφέραμε βέβαια σε όλα τα σημεία, αλλά η αρχική μας θέση ήταν αυτή. Είναι ένα θέμα, επαναλαμβάνω, στο οποίο πετύχαμε αρκετή συνένεση. Η πρόσφατη ιστορία αποδεικνύει πως οι καταγγέλλοντες έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν και υπάρχει ένα νομικό κενό στα περισσότερα κράτη-μέλη και γι' αυτό είναι σημαντική αυτή η οδηγία η οποία έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτό το κενό. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια επίμαχα ζητήματα, αλλά νομίζω πως τελικά καταλήξαμε σε μια διατύπωση η οποία, επαναλαμβάνω, βρίσκει τους περισσότερους σύμφωνους. Το πιο επίμαχο θέμα είναι το σχετικό με την ιεραρχία. Δηλαδή, τι εννοώ, μέχρι ποιο βαθμό το εξωτερικό κανάλι καταγγελίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πότε εξαντλούνται οι εσωτερικοί διάβλοι καταγγελίας. Δηλαδή, όταν δεν, ε, η εσωτερική οδός καταγγελίας δεν προσφέρει επαρκή εχέγγυα ασφάλειας. Να σας πω λοιπόν στο κείμενο στο οποίο καταλήξαμε ε, οδηγεί στο εξή. Θα πρέπει καταρχήν στο εσωτερικό των επιχειρήσεων να προσπαθούμε να δώσουμε μια λύση σε αυτό το θέμα, αλλά να αναγνωρίζουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις αυτό δεν είναι δυνατόν. Και θα πρέπει να δώσουμε κάποιες εξασφαλίσεις στους καταγγέλλοντες, έτσι ώστε να μπορούν να επιλέξουν την οδό καταγγελίας η οποία θα είναι η πιο αποτελεσματική χωρίς να χρειαστεί να δικαιολογήσει με πολύ λεπτομερή τρόπο ε, κάθε βήμα που έκανε γιατί δεν επέλεξε για παράδειγμα την ε, εσωτερική δίωδο καταγγελίας και τα λοιπά. Τα υπόλοιπα επίμαχα ήταν η ανωνυμία και η προστασία ε, της ταυτότητας. Εμείς δεν πετύχαμε εδώ συμφωνία, αλλά είναι σημαντικό οι πλατφόρμες οι οποίες συλλέγουν αυτές τις καταγγελίες θα πρέπει να εξασφαλίζουν το απόρριτο. Και θεωρούμε πως αυτό είναι ένα σημείο κλειδί. Στα πλαίσια της οδηγίας ακούσαμε προτάσεις όλων των ειδών. Μιλήσαμε για ένα μεγάλο κατάλογο, ο οποίος τελικά μειώθηκε και έχουμε τώρα πιο συγκεκριμένες διατάξεις Ε, και βεβαίως περιοριστήκαμε στα όσα είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής μας. Δεν επεκταθήκαμε σε άλλα χωράφια. Προσπαθήσαμε να ξεκαθαρίσουμε το τι γίνεται με τις υλικέ απαιτήσει των καταγγελόντων και πώς μπορεί να γίνει δικαιούχος αυτής της οδηγίας σε επίπεδο προστασίας και τις διατάξεις τι οποίε θα πρέπει μετά τα εθνικά κοινοβούλια να διατυπώσουν και να ψηφίσουν. Αυτά ήταν τα βασικά στη συζήτηση που κάναμε. Θεωρούμε πως καταφέραμε να πετύχουμε τη συνένεση ε, δεδομένης της ε, πολυγλωσσίας ε, αυτής της αίθουσας. Βεβαίως υπάρχουν σημεία στα οποία δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, αλλά θεωρώ πως γενικά τα πήγαμε καλά. Ευχαριστώ όλους τους σκιώδεις και όσους συμμετείχαν άμεσα ή έμεσα στη σύνταξη του κειμένου. Ε, Ευχαριστώ Μιγγέλ, γι' αυτό πάμε στις ομάδες. Ο Βεν Λάγκεν, εκ μέρους του ΕΛΚ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Δεν ε, μπορώ να συμμεριστώ την αισιοδοξία του εισηγητή. Δεν είχαμε καθόλου χρόνο να συζητήσουμε τις συμβαστικές. Δεν είχαμε συνάντηση των ε, σκιωδών εισηγητών. Ήταν πράσινη εβδομάδα Οπότε ο συνάλφος που λέει τώρα ότι κατέβαλε κάθε προσπάθεια, ε, απλά δεν ισχύει αυτό. Δεν συζητήθηκαν οι τροπολογίες μας, ούτε λήφθησαν υπόψη. Αυτό θεωρώ το λογικότερο ήταν να αναβάλουμε την απόφαση για την επόμενη συνεδρίαση για να μπορέσουμε να συζητήσουμε κάποιες συμβιβαστικές λύσεις. Αυτή είναι η πρότασή μου. Εάν επιμένει στην ψηφοφορία ο εισηγητής, έχουμε εμείς έξι σημεία στα οποία θα καταψηφίσουμε να τα συνοψίσω. Όλοι συμφωνούμε ε, μετά την Εξεταστική Επιτροπή για τον Παναμά. Συμφωνούμε και μετά τις αποφάσεις στο Λουξεμβούργο πως απαιτείται μεγαλύτερη προστασία. Αλλά όταν ζητάνε απόλυτη ανωνυμία του πληροφοριοδότη πράσινη και σοσιαλδημοκρατία, ε, δεν χρειάζεται άλλη προστασία. Πρέπει να υπάρχει ε, μια δυνατότητα. Δηλαδή η προστασία έχει νόημα όταν δεν υπάρχει ανωνυμία. Αλλιώς δεν στέκει. Να αναφέρω κάτι άλλο. Οι τρόποι καταγγελίας. Εάν πρέπει να γίνει καταγγελία αρχές, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι καταγγελίας. Εξού και η ιεραρχία που πρότεινε η Κομισιόνα, η οποία κατά την απόψή μας είναι το σωστό. Κατόπιν ε, το θέμα των ασαφών διατυπώσεων. Παραδείγματος χάρη η 57 η τροπολογία particularly λέει εδώ πέρα. αυτό δηλαδή σημαίνει και οτιδήποτε άλλο. Και βεβαίως ε, θα έπρεπε ίσως να το συζητήσουμε κατόπιν η δυνατότητα που μας δίνει ο εισηγητής τι λέει εδώ πέρα, αν υπάρχει μία έκθεση θα μπορεί να την, να την διορθώσει ο καταγγέλων. Τι είναι αυτό, τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Μετά το βάρος της ε, αποδείξεως. Για αυτόν ο οποίος ε, δίνει τις πληροφορίες. Ε, δηλαδή έχουμε φτάσει σχεδόν στο καθεστώς της ε, Στάζη που είχε πληροφορίες ε, για τους πάντες. Έχουμε λοιπόν αυτά τα έξι σημεία στα οποία είχαμε προτείνει τις ε, συμβαστικές προτάσεις. Όπως σας είπα το λογικό τώρα είναι να αναβληθεί η ψηφοφορία για να μην καταλήξουμε σε αρνητική ψήφο. Ωραία, Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Για τους σοσιαλδημοκράτε, ο κ. Σκοφότ. Ευχαριστώ. Να πω ότι η ομάδα του SND καλωσορίζει θερμά την πρόταση Ευρωπαϊκή Επίτροπή, Είναι μια πρόταση που ζητούσαμε επί καιρών. Από το LuxLeaks στα Panama Papers, μετά στα, στα διάφορα στο Danske Bank κλπ. Στο ξέπλυμα χρήματο, είχαν πολλά σκάνδαλα που ήρθαν στο φω χάρη στου πληροφοριοδότε αλλά η προστασία αυτών που παρέχουν πληροφορίε, παραμένει ανεπαρκέστατη στην Ευρώπη. Με την έγκριση και την εξέταση αυτού του θέματο, βελτιώνουμε την κατάσταση. Το S&D έχει εισαγάγει νέα άρθρα όσον αφορά τι υποχρεώσει των κρατών μελών να συνεργαστούν μεταξύ του. μέσω του ΤΑΚΣ, του τάξ του, του ΠΑΝΑ, αποκαλύψαμε ότι οι αρχέ των κρατών μελών δεν συνεργάζονται επαρκώ με αποτελεσματικό και ανοιχτό τρόπο με τις νέες διατάξεις που με τα χαράς βλέπουμε να συμπεριλαμβάνεται στις συμβαστικές τροπολογίες θα γίνεται μια πραγματική συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και αυτό γίνεται μια προϋπόθεση νομική και θα πρέπει τα συστήματα υποβολή καταγγελιών να εξασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που παρέχουν οι πληροφοριδότε και θα πρέπει να ξέρουμε και ποιο έχει πρόσβαση πληροφορίε και πότε, ώστε παρά μόνο αυτοί ε, που έχουν το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση στο εμπιστευτικό ε, αυτό υλικό και θα προστατεύουμε την ταυτότητα και την ε, ζωή αυτών των πληροφοριωτών. Λοιπόν, με προθεσμία μιας εβδομάδας για να παρασχεθεί σημείωμα αποδοχής και ένα μήνα για μια πρώτη απάντηση που θα δοθεί σε εκείνο που δίνει τις πληροφορίες. Αυτά είναι τα όρια που έχουν τεθεί εμείς αυτό θέλαμε, αλλά οι άλλες ε, ομάδες δεν συμφωνούσαν, δεν πετύχαμε τη σωστή πλειοψηφία. Συγχαίρουμε τον εισηγητή για τη δουλειά που έκανε. Προσβλέπουμε σε έγκριση κατεπηγόντος του κειμένου αυτού, που είναι απαραίτητο για τους καταγγέλλοντες στην Ευρώπη και θέλουμε η διαδικασία να είναι καλύτερη και όπως είπε και ο Βέρνε Λάγκεν, θα θέλαμε ε, να είχε ακολουθηθεί μια καλύτερη διαδικασία στην όλη αυτή υπόθεση. Ευχαριστώ, ECR, ο θα μιλήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Προσπάθησα να πετύχει τη σωστή ισορροπία. Αλλά οι πολλές τροπολογίες, οι 183 τροπολογίες, δείχνουν ότι υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις όσον αφορά τον τρόπο που προστατεύονται οι πληροφοριοδότες και σε ποιο βαθμό θα πρέπει να παραμείνουμε στις αρμοδιότητες της Επιτροπής μας, εφόσον αυτή είναι μια γνωμοδότηση. Πρωταρχικά πρέπει να επικεντρωθούμε επί οικονομικών ε, και χρηματοστατικών πτυχών των υποθέσεων αυτών. Η ομάδα μας θεωρεί ότι οι διαδικασίες για εσωτερικούς διάβλους υποβολής καταγγελιών προτείνεται να καταργηθούν και θα πρέπει να υπάρχει μια προσέγγιση κατά περίπτωση πιστεύουμε. Χαίρομαι που τροπολογίε μου για εξαιρέσει για τι καταγγελίε. δεν θα πρέπει να ισχύουν μόνο για τι ιδιωτικέ επιχειρήσει, αλλά και αυτέ που είναι πολύ στενά συνδεδεμένε με τα χρηματοπιστωτικά. Πρέπει να προστατεύονται οι καταγγέλλοντε, να στηρίζονται, αλλά βλέποντα την πρόοδο που ακολουθεί αυτή η γνωμοδότηση, προτείνω στην ομάδα μα αποχή. βλέποντα εξελίξεις που πάνω σε αυτό το θέμα, προτείνω αποχή στην ομάδα μου. Ευχαριστώ κύριε Ζέλα δεν έχουμε κάποιον από την Άλτε. Μπορούμε να επιστρέψουμε λοιπόν στον εισηγητή. Α, συγγνώμη. Μόλι. Μόνο ένα λεπτό. Εντάξει, θα κάνω ό,τι μπορώ. Να ευχαριστήσω και εγώ τον Μιγγέλ για τη δουλειά που έκανε και πάνω σε αυτά που είπε ο ο Λάγκερ. Ε, είμαστε περιορισμένοι χρονικά, δεν είχαμε επαρκή χρόνο για δελεχή συζητήσει, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, διότι θα έπρεπε να απολυθεί και αλλού η γνωμοδότηση. Χαιρόμαστε που παρουσιάστηκαν αυτέ οι τροπολογίε συμβαστικέ πλευρά συζητητού. Να πρέπει να γίνεται όμω στον τόπο εργασία αυτή η παροχή πληροφοριών, αλλά οπουδήποτε εργάζεται κανεί, στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, θα πρέπει να ε, ε υπάρχει κατάλληλη προστασία. Συμφωνούμε για διάβλου ε, καταγγελιών. Θα πρέπει οι πληροφοριοδότες καταρχάς εσωτερικά να κάνουν καταγγελίες, αν αυτό είναι ανέφικτο. Θα πρέπει ίσως να κάνουν τι καταγγελίες έξω από το όριο αυτό. Πρέπει να προστατεύονται από οι καταγγέλλοντε. Ξέρουμε ότι πολύ συχνά οι καταγγέλλοντε ε, τιμωρήθηκαν. Ε, ακολουθήθηκε τιμωρητική δράση εναντίον αυτών και των οικογενειών τους. Άρα γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ανωνύμων ε, καταγγελιών εμπιστευτικού χαρακτήρα, επευλήθησαν τροπολογίε για την ενημέρωση των πληροφοριοδοτών, γιατί πολύ συχνά παραμένουν στο σκοτάδι για κρίσιμε πληροφορίε που σχετίζονται για το πώ χρησιμοποιούνται οι πληροφορίε που διέθεσαν. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε σε περίπου μία ώρα πάνω σε αυτό και είναι κρίμα που δεν είχαμε το χρόνο να ψηφίσουμε, να το συζητήσουμε επαρκώ, αλλά είναι σημαντικό το ότι έλθει να το στηρίξει. Όπω υπόθηκε πριν, υπάρχει ευρία υποστήριξη για αυτά που κάνουμε και θα ήταν κρίμα αν τελικά έδειχναν ότι είναι στην αντίθετη πλευρά από, αυτό που θα έπρεπε να, από αυτή που θα έπρεπε να είναι. Ευχαριστώ. Τώρα θα δώσουμε το λόγο λοιπόν στον εισηγητή. Θα είμαι πάρα πολύ γρήγορος και να σας πω πως είναι προφανές πως το χρονοδιάγραμμα δεν ήταν ευνοϊκό και δεν μπορέσαμε να κάνουμε συναντήσεις με τους σκιώδες για τους λόγους που εξήγησα. Και θα ήθελα να τονίσω το εξής. Θα πρέπει να σταθούμε στο ύψος των προσδοκιών των συμπολιτών μας. Όλοι θυμούνται τα άτομα που πέθαναν σε τραγικές συνθήκες Και αυτά τα γεγονότα μας οδηγούν στο να δράσουμε χωρίς καμία καθυστέρηση. Μιλάμε εδώ για μια οδηγία η οποία έχει ευρύ πεδίο. Η στήριξη αυτής της οδηγίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα στείλει ένα ηχηρό μήνυμα και παράλληλα δίνει περιθώριο στα κράτη-μέλη να μπορούν να προσαρμόσουν ε, στις δικές τους συνθήκες τα κείμενα αυτά. Υπάρχει ένα νομικό κενό και θα πρέπει να το καλύψουμε. Ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα με τη σειρά μου και εγώ να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Ο Μπέρναρτ. Θα ήθελα να παρακαλέσω ακόμη μία φορά να αναβληθεί η ψηφοφορία γιατί δεν είχαμε την δυνατότητα να συζητήσουμε για τις συμβιβαστικές και να βρεθεί μία λύση. Αυτό ζητάω, να πάει στην επόμενη συνεδρίαση. Έχουμε χρόνο. Thank you. Uh, I understand that uh, as often unfortunately happens uh... Ε, ευχαριστώ. Αντιλαμβάνομαι ότι όπω συμβαίνει συχνά δυστυχώ έχουμε θέματα χρόνο διαγράμματο τα οποία μα επιβάλλει η κατά κύριο λόγο αρμόδια επιτροπή, οπότε δεν έχει νόημα να ψήσουμε μια γνωμοδότηση πάρα πολύ αργά. Γι' αυτό φοβάμαι ότι πρέπει να περάσουμε να ψήσουμε τους ή Πρέπει να διακόψουμε θα περάσουμε τις ψηφοφορίες. Ωραία. Να κάνουμε λοιπόν μια δοκιμή, μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Όλοι σας παρακαλώ πολύ βγάλτε τις κάρτες σας και θα κάνουμε μια δοκιμή να δούμε αν λειτουργούν. τρία μέλη, δύο μέλη. Α, ωραία. Εντάξει, τώρα έχουμε ένα παραπάνω. Ωραία, τελείωσε η δοκιμή. Θα ξεκινήσουμε με την πρώτη ψηφοφορία. Είναι τα, οι απαιτήσει προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων, Φέρμπερ Μάρκους, συμβιβαστική M κατά αποχές εγκρίνεται. Εν υπέρ κατά εγκρίνεται. Ο εγκρίνεται. Εννέα υπέρ κατά για να δούμε την εννιά. άρχεται η ψηφοφορία λίγη εγκρίνεται. Π. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική A υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. B υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. E υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. FA υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. GA υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. H Α, περάσαμε το GA, συγγνώμη. Όχι, δεν ψηφίσαμε τη G. Λοιπόν, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. GA υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία. Έχουμε μία προφορική τροπολογία που έχουν ζητήσει οι πράσινοι. Έχετε εσείς αντίρρηση? Πρέπει να υπάρχει παρκής αριθμός, ναι. Θέλουμε να τονίσουμε πως υπήρχε χρόνος και δεν νομίζω ότι είναι ε, λόγος που το ζητάτε προφορικά. Είχατε χρόνο και θα πρέπει να το έχετε κάνει γραπτά. Το I λοιπόν, συμβαστική I λέει ο πρώτος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική K υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Q με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λοιπόν, όπως τροποποιήθηκε, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Α, σήμερα δεν τα πάω καλά. Και ξέρετε γιατί γιατί τα έχουν κάνει άλλο χρώμα. Γιατί έχετε αυτά τα γκρίζα και αυτά τα αλφα. Όχι, να γυρίσουμε στο κάνω όπως το κάναμε παλιά. Να μην μπερδεύομαι. Εν πάση περιπτώσει, 37 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά ελέγχουμε την 53 παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. 23-18. 54 υπέρ. Κατά. Ποχές. Απορρίπτεται. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται με την ίδια πλειοψηφία, αλλά αν θέλετε μπορούμε να το δούμε και ηλεκτρονικά. Θέλετε? Ωραία. Ηλεκτρονικά λοιπόν άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 22-19. 56. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και τώρα λοιπόν, όπως τροποποιήθηκε ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Άλλος ένας συνάδελφος πρέπει να ψηφίσει, πέρας 33 υπέρ, 8 ε, κατά, άρα λοιπόν, ε, εντάξει, για το επόμενο λοιπόν ε, μπορούμε να ξεκινήσουμε με την ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας, 34 υπέρ, 8 κατά, 0 αποχές. Λοιπόν, οπότε μπορούμε να συγχαρούμε τον εισήγητη και να περάσουμε στο δεύτερο κομμάτι. Προληπτική εποπτεία επενδυτικών εταιριών, ανθρωπολογία 30. Α, καταπίπτει, μάλιστα. Περνάμε λοιπόν συμβαστική Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 15 γιουρ υπέρ υπέρ, ναι, κατά αποχές εγκρίνεται, 16 γιουρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική σ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, γιούρι 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, γιούρι 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, γιούρι 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, Γιούρι 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, Γιούρι 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, Γιούρι 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, Συμβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, Τροπολογία 53 υπέρ κατά, δεν βλέπω τους πράσινους, έχει τα θέση επί του θέματος. Α, όχι. Μάλιστα. Να την επαληθεύσουμε λοιπόν, να έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 22 εναντί 20. Καταπίπτει. Περνάμε στην ε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική I υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική που είμαστε σελίδα 8. IA υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική και υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 179 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 180 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 181 υπέρ κατά να την επαληθεύσουμε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 23 υπέρ, 21 κατά, 182 υπέρ. Κατά. Η από εδώ πλευρά δεν σηκώνει χέρια. Λοιπόν, να το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 22 με 16. Γιούρι 50 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 193 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 194 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική M υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, γιούρι 51 υπέρ κατά να την επαληθεύσουμε, άρχεται η ψηφοφορία. Να δούμε. Πέρας. Εγκρίνεται 24 έναντι 16. Συμβαστική N υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική O υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική P υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Γιούρι 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Γιούρι 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 και 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, Γιούρι 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, Γιούρι 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 6 υπέρ, Γιούρι 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 1 και 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται, 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται, Γιούρι 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται, Γιούρι 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται, 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται, Γιούρι 9 υπέρ κατά αποχές, να την απολυθεύσουμε, την 9 της Γιούρι. Πέρας, η ισοψηφία απορρίπτεται λοιπόν. Γιούρι 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Γιούρι 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Γιούρι 12 είναι ταυτόσημη, ναι. 23 λοιπόν υπέρ κατά άλτε μάλιστα. Άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν. Δεν καταλαβαίνω. Ναι. Πέρας. Η ισοψηφία απορρίπτεται. Καλά κάναμε λοιπόν και το επαληθεύσαμε. Η 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 25 καταπίπτει, άρα πάμε στην 3 και 26 καταπίπτει, 27 υπέρ, κατά να την επαληθεύσουμε, άρχεται την ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται Γιούρι 13 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 28 υπέρ κατά να την επαληθεύσουμε. Λοιπόν, άρχεται τη ψηφοφορία για το 28. Πέρας. Απορρίπτεται. 23-29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική R υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά να την επαληθεύσουμε. Την 4 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την πρόταση της Κομισιόν όπως τροποποιήθηκε. Με ονομαστική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. 25 υπέρ, 9 κατά, καμία αποχή. Η απόφαση για διοργανικές διαπραγματεύσεις, άρχεται η ψηφοφορία, ονομαστική. Πέρας. 35 υπέρ, 9 κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια λοιπόν στην εισηγήτρια. Περνάμε τώρα στο σχέδιο γνωμοδότησης για τα πλαστικά. Η Μπάρμπαρα Κάπελ είναι η συγγήτρια. Συμβιβαστική Α, υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος. Πιστεύω ότι εγκρίνεται όμως. Ας ελέγξουμε να δούμε τη διαφορά των ψήφων. Πέρας. 4 υπέρ, 10 ψήφοι κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 86 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι απορρίπτεται με την ίδια 87 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αποσύρεται 88 τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 89 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 90 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Α, 92. 92 υπέρ. 92. Πάμε πίσω στην 92 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 20 ψηφίσαμε. Ψηφίσαμε την 20. Μπορώ να επαναλάβουμε. Την ψηφίσαμε. Γιατί ξέχασα την 29. Λοιπόν, 20 ξανά. Απεσύρθη 93. Στον κατάλογό μας έχει αποσυρθεί 93. Έχει αποσυρθεί λοιπόν. Η 93 αποσύρεται. Ψηφίζουμε την 20. Κάποιος ζήτησε να ξαναψηφίσουμε. Και από εδώ, την γραμματεία. Λοιπόν, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική D δεν υφίσταται πλέον προφορική τροπολογία που αφορά το άρθρο 7α νέο. Τροπολογία 94, προφορική τροπολογία, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το πρωτότυπο κείμενο 94, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 95, υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία για την 95. Πέρας. Εγκρίνεται. 96. Πρέπει να ψηφιστεί. 96 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 97 υπέρ. Κατά. Έλεγχος για την 97. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 98 υπέρ κατά άποχες σε υπέρ έλεγχος για την 98 άρχεται η ψηφοφορία Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 99 υπέρ. Κατά. Έλεγχος για την 99. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ισοψηφία άρα απορρίπτεται. 21-21. 100 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 103 υπέρ κατά έλεγχος νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά ελέγχουμε Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 105 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 104 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική F υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 22. Πού είναι. 22 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 108 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος για την 108. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 109 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 23 και 110 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται θα έλεγα 27 υπέρ κατά αποχές αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 112 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 114, έτσι. 114 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική I υπέρ. Η Άλντε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 118 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ένα υπέρ, κατά, δεν βλέπω χέρια για την ένα. Κάνουμε ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Οι 119 και 120 έχουν αποσυρθεί, λέει ο πρόεδρος. Συγγνώμη. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική J υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 43 υπέρ κατά έλεγχος γιατί 43 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται συμβαστική κάπα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 52 υπέρ κατά έλεγχος για την 52 άρχεται η ψηφοφορία. πέρας εγκρίνεται 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική νη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται συμβαστική ο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 υπέρ κατά Έλεγχος για την 60, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 22, 20, 61 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 62 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 63 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική π υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την πρώτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που τροποποιήθηκε ονομαστική ψηφοφορία που άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. 25 ψήφοι υπέρ, 19 κατά, μια αποχή. Εγκρίνεται συγχαρητήρια λοιπόν στον εισηγητή και το σχέδιο γνωμοδοτήσεως για τους πληροφοριοδότες Μιγγέλ Βιέγκας. Συμβαστική ανθαϊπέρ κατά αρχές έλεγχος άρχεται. Πέρας εγκρίνεται συμβαστική β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική ε υπέρ κατά δεν βλέπω το έλεγχος για την ε, έτσι, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 26-19 συμβαστική F υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται συμβαστική G υπέρ κατά έλεγχος για τη συμβαστική G άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 2318 H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. I υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 171 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εγκρίνεται, αλλά αυτό θα το ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 22-15 με 8 αποχές, συμβαστική και υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, L υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 193 υπέρ, κατά Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ισοψηφία, άρα λοιπόν απορρίπτεται 21 και 21. M, συμβαστική υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 201 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 205 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 206 υπέρ κατά τα αποχές 206 ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία 206 τροπολογία 206 πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 23-20 22 υπέρ κατά αποχές και πάλι ηλεκτρονικά Νομίζω έχει υπερψηφιστεί, αλλά θέλω να το δούμε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Και εδώ πάλι έχουμε ισοψηφία 22 με 22 απορρίπτεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικά και πάλι την 23 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Αποχές 22-19. Εν. Συμβιβαστική εν. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονικά την 27 παρακαλώ άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 25-17 ο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Π υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πρώτη υπέρ Υπορθμόν 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ κατά ηλεκτρονικά παρακαλώ την 38. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ κατά τη 40 παρακαλώ ηλεκτρονικά πέρας απορρίπτεται 23-21 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 υπέρ κατά 42 ηλεκτρονικά παρακαλώ Πέρας. Απορρίπτεται. 23-21. 43. Υπέρ κατά αποχές. Ελκ για, την, για τη 43. Ελκ είστε κατά. Απορρίπτεται. 45. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ κατά Διαστηκά, γιατί 46 ηλεκτρονικά παρακαλώ άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται λοιπόν. Πέρας ψηφοφορίας έχει εγκριθεί 29 με 12. 47 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ κατά αποχές. Για να δούμε τη 49. Λοιπόν, είδα να εγκρίνεται, αλλά στο δούμε και ηλεκτρονικά. 33, 10, 50. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 51. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52. Καταπίπτει. 53. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 54. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 55. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 56 υπέρ Γκου, είστε υπέρ της 56 κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 60 υπέρ κατά αυτό θα το δούμε και ηλεκτρονικά, γιατί βλέπω κάποιους να έχουν μετακινηθεί μέσα στις ομάδες, ίσως πρόκειται και για σφάλμα. Ηλεκτρονικά λοιπόν, πέρας ψηφοφορίες, απορρίπτεται. 22 με 21. 58 και 59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 61 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 75 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται και μετά από την 76 μέχρι την 83 όλες μαζί. Όχι, η 76 ξεχωριστά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα 77 με 83 υπέρ κατά Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Vote is closed. Rejected. 20... λοιπον λοιπόν 23-21 και περάμε τώρα στην 85 υπέρ κατά ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 24 με 21, 87 μέχρι την 90, όλες μαζί υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 4 και 91 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 92 υπέρ, κατά, ηλεκτρονικά την 92 παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 5 και 93 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 95 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Όλες μαζί 96 με 102 αν συμφωνείτε μέχρι τις 100, 96 με 100 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 102 Α, 100 με 102. Όχι, η 100 ήταν με τις προηγούμενες που ψηφίσαμε όλες μαζί. Ωραία, να ψηφίσουμε και την 100 για την 100 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται οι 101 και 102 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Για το κείμενο ολόκληρο, έτσι όπως τροποποιήθηκε, ονομασική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 24 υπέρ, 15 κατά εγκρίνεται συγχαρητήρια στον εισηγητή. Now I will pass the Τώρα θα δώσω την Προεδρία και πάλι για την κοινή μας συνεδρίαση με την Επιτροπή Γυναικών. Σας ευχαριστώ.